Αγαπητοί συνάδελφοι, σας προτείνω να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ πολύ να μας συγχωρήσετε για την καθυστέρηση, αλλά ε, κάναμε κάποιες αλλαγές ε, στην ημερήσια διάταξη και αυτό προκάλεσε την ε, καθυστέρηση. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν. Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε στην συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού. Θα ξεκινήσουμε με την έγκριση της ημερησίας διατάξεως. Να σας πω ότι προέκυψαν κάποιες δυσκολίες Οι ε, νεαροί ε, του βραβείου Καρλομάγνος ε, κάνουν κάποια φωτογράφηση και δεν είναι ακόμα εδώ. Και η κυρία Τρίπελ, η οποία θα έπρεπε να μας μιλήσει για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι λόγω κίνησης ακόμα στους δρόμους. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την έκδοση Μακοβέη και να προχωρήσουμε μετά στην παρουσίαση του βραβείου Καρλομάγνους και μετά να συνεχίσουμε με την κανονική μας ημερήσια διάταξη έτσι όπως ε, ε, την έχετε ήδη μπροστά σας. Ε, σας ζητώ λοιπόν κατανόηση. Έχετε σχόλια όσον αφορά την ημερήσια διάταξη, όχι από ό,τι φαίνεται και επομένως εγκρίνεται η ημερησία διάταξη. Σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών. Έχουμε τα πρακτικά ε, του Οκτωβρίου, των συνεδριάσεων της Επιτροπής μας του Οκτωβρίου. Έχετε επ' αυτών σχόλια? Όχι από ό,τι φαίνεται. Και επομένως προτείνω όσοι ήθιστε να θεωρήσουμε τα πρακτικά ε, ως ε, αποδεκτά. Σημείο 3. Ανακοινώσεις της Προέδρου. να σας μιλήσω για το γλωσσικό καθεστώς. Έχουμε διάφορες γλώσσες, μεταξύ των οποίων τα ελληνικά. Μπορείτε να μιλήσετε και να ακούσετε ελληνικά. Απαριθμεί τις γλώσσες η Πρόεδρος. Ε, σχετικά με την πρωτοβουλία ε, για την απασχόληση των νέων στα κράτη-μέλη. Η είναι ο συνάδελφός μας, ε, κύριος Νεκόβ Μομτσίλ. Κύριε Μομτσίλ, θέλετε να πάρετε τον λόγο. Όχι, επομένως μπορούμε να περάσουμε απευθείας εις τις ψηφοφορίες. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Με συγγνώμη 9, διορθώνει η πρόεδρος, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές ε, καλύτερα να επαληθεύσουμε το αποτέλεσμα Ξαναψηφίζουμε λοιπόν με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 13 ψήφοι υπέρ, 14 ψήφοι κατά. Τροπολογία 15. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές. Ε, καλύτερα να ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά ελέγχουμε λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Με 14 ψήφους κατά. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές δεν είμαι σίγουρη. Η Ηλεκτρονική επαλήθευση νομίζω ότι θα έχουμε την ίδια πλειοψηφία αλλά καλύτερα να ψηφίσουμε ξανά επί της 19 πέρας της ψηφοφορίας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 Πέρας της ψηφοφορίας. 14 ψήφοι κατά, 13 ψήφοι υπέρ, απορρίπτεται. Τροπολογία 27 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές Νομίζω πως έχει απορριφθεί, αλλά προτιμώ να το ελέγξουμε. Τροπολογία 29, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 14 ψήφοι είναι κατά, 12 υπέρ, επομένως απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. αποχεσε εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά. αποχεσε εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά. Αποχές Νομίζω πως απερίφθη, αλλά θα ήθελα να το ελέγξουμε τροπολογία 33 άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας απερίφθη 10 ψήφοι μάλλον 11 γιατί μετράμε και αυτό που δεν έχει την κάρτα του 17 κατά 34 ε, υπέρ κατά αποχές επαλήθευση Ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν. Νομίζω ότι δεν ψήφισε καλά η σοσιαλιστική ομάδα, δεν σήκωσε τα χέρια της. Πέρας της ψηφοφορίας. Λοιπόν, 14 ψήφοι υπέρ. Όχι, διορθώνω λέει η Πρόεδρος. 14 ψήφοι κατά, 13 ψήφοι υπέρ. Άρα απερίφθη. Ε, μάλλον δεν λειτουργήσε καλά το μηχάνημα της ε, Σιλβία από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, 35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τέλος, Ε, τελευταία ψηφοφορία άρχεται με ηλεκτρονική ψηφοφορία πέρας 26 ψήφοι υπέρ ε, καμία ψήφος ε, εναντίον μία αποχή και επομένως με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε και ευχαριστούμε και συγχαίρομαι τον συνάδελφο Νεκόβ Μομτσίλα Λοιπόν, συνεχίζουμε την ημερήσια διάταξη, αλλά όχι με τη σειρά της, διότι η συγγήτρια του σημείου 6 δυστυχώς είναι μπλοκαρισμένη σε ένα τρένο. Ε, ούτε το σημείο 7 μπορούμε να δούμε, διότι οι νικτές του βραβείου ε, Σαρλεμάνι ε, βγάζουν φωτογραφίες με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, αλλά έχουμε εδώ το συνάδελφο Μαλτέζε, οπότε μπορούμε Οπότε μπορούμε να ε, ξεκινήσουμε ε, με τον πλουραλισμό στα μέσα ε, ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάσει του άρθρου 54 έχουμε τη διαδικασία μας. Η συγητής είναι ο κύριος Κούρτσιο Μαλτέζε. Ε, είχα ήδη αναφέρει το άρθρο 54 λοιπόν. Είμαστε αρμόδιοι όσον αφορά τα θέματα ε, μέσων ενημέρωσης. Κύριε Κούρτσιο, σας δίνω το λόγο. Έχετε πέντε λεπτά για να μας παρουσιάσετε το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ίσως δεν θα μου πάρει ούτε καν πέντε λεπτά. Η φιλοσοφία Ε, μάλλον να, ξεκινήσω όταν θα έχουν σταματήσει τα πηγαδάκια γιατί δεν μπορώ έτσι. Λέει ο κύριος Μαλτέζε. Bene. Mm, ο κύριος ε, Κούρσιο Μαλτέζε. Εγώ ξεκίνησα από την δικιά μου ε, εμπειρία. Ε, ποτέ δεν στην καριέρα μου ως δημοσιογράφος δεν είχα ε, συναντήσει έτσι μία αντιμετωπίσει μια αντιμετωπίση μια κρίσιμη περίοδο. Το είπε και η Πρόεδρος ε, πριν, το θέμα της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ. Εγώ προσπάθησα να κάνω μια σύνθεση των πιο ουσιαστικών στοιχείων με τρόπο όμως σαφή ε, και απλό έτσι ώστε να δώσω ένα ε, συνολικό πλαίσιο κατά κάποιο τρόπο της δυνατότητας δράσης ε, και να καταδείξω τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά την πληροφόρηση, διατρέχουμε τον κίνδυνο να επικεντρωθούμε μονάχα ε, στις ε, τροποποιήσεις των τελευταίων χρόνων που είναι βεβαίως ε, το φαινόμενο των fake news, των ψευδών ειδήσεων και σε ορισμένες χώρες και για ορισμένες περιπτώσεις βεβαίως παραβιάσεις της ελευθεροτυπίας και της ελευθερίας έκφρασης που είναι κάτι εξαιρετικά σοβαρό. Εγώ αναφέρθηκα σε ε, όλα τα θέματα αυτά. Αναφέρθηκα επίσης στην ε, ανάδυση ε, πολλών δύσκολων και επικίνδυνων περιπτώσεων όπως ας πούμε την δολοφονία της συναδέλφου στην Μάλτα που αποτελούν κατά κάποιο τρόπο ένδειξη αλλαγών που έχουν επέλθει, επικίνδυνων αλλαγών που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια. Αυτό που με απασχολούσε όμως ιδιαίτερος είναι να δώσω ένα γενικό γενικότερο πλαίσιο των μέσων μαζικής ενημέρωσης που τα τελευταία 200 χρόνια, τους δύο τελευταίους αιώνες, ε, ακολουθούν την πορεία της ε, κοινωνίας αυτό που έλειψε τα τελευταία χρόνια είναι ε, η κοινωνική διασύνδεση πέρα από την οικονομική ε, της ε, κοινής, ανάμεσα στην κοινή γνώμη και τον κόσμο των δημοσιογράφων, των επαγγελματιών δηλαδή του, του κλάδου. Ε, γιατί η ελεύθερη ε, είδηση και η ελεύθερη ε, πολύφωνη έκφραση της ελευθερίας έπρεπε να χρηματοδοτείται από τον ίδιο τον κόσμο, από το, από το κοινό. Αυτό όμως τα τελευταία χρόνια έπαψε να ισχύει μέσα από τη συγκέντρωση στα χέρια των ολίγων της δύναμης του να ακουστεί η φωνή ή το να γίνει ε, η διαφήμιση και επομένως όλο και πιο συχνά ε, η ενημέρωση λειτουργεί με τρόπο χειραγωγικό Ε, εγώ ανέφερα ότι η υπερβολική συγκέντρωση στα χέρια ολίγων των μέσων ενημέρωσης ε, είναι κάτι επικίνδυνο και πρέπει να μας απασχολήσει γιατί ε, αυτοί οι λίγοι παίχτες στον τομέα των μέσων ενημέρωσης που πολλές φορές δεν είναι καν Ευρωπαίοι 90% ας πούμε των υπεύθυνων και των δημοσιεύσεων ε, ε, διαφημίσεων ή ε, διαφημίσεων είναι στα χέρια μη ευρωπαϊκών εταιριών και επομένως δυσκολεύει πάρα πολύ η κατάσταση και για τους εκδότες και για τις ευρωπαϊκές ομάδες ή εταιρείες ενημέρωσης και για τους ίδιους τους δημοσιογράφους. Τέλος, οι συνθήκες εργασίας ε, οι οποίες είναι ε, όλο και πιο ε, ασταθείς κυρίως για τους νέους δημοσιογράφους είναι κάτι που μας απασχολεί ιδιαιτέρως. Έχουν ιδιαίτερα ε, δυσκολέψει οι συνθήκες και έχουν γίνει πολύ χειρότερες. Ε, έχει επιδεινωθεί ε, και το θέμα των μισθών των νέων δημοσιογράφων αλλά και οι δυνατότητες κατάρτισης που έχουν. Αυτά είναι τα κεντρικά στοιχεία τα οποία προσπάθησα να αναλύσω έτσι ώστε να διαγράψω έτσι ένα πλαίσιο πλαίσιο των αιτίων που οδηγούν ε, σε αυτήν ε, ε, την δύσκολη κατάσταση των fake news αλλά και του ιδιαίτερα χαμηλού ποιοτικού επίπεδου της πληροφόρησης. Αυτά τα θέματα νομίζω ότι μας απασχολούν πάρα πολύ στην Επιτροπή μας και επομένως ε, περιμένω να ακούσω πολλές νέες ιδέες και από εσά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα τώρα πρώτα να παρακαλέσω να λάβουν το λόγο οι σκιώδεις εισηγητές και θα αρχίσω με τον κύριο Νέκοφ ο οποίος εκπροσωπεί τον σκιώδη εισηγητή Τράγκητσι. Ευχαριστώ. Θα σας παρουσιάσω την θέση του κ. Τραγκίτσε, ο οποίος θεωρεί καλή την έκθεση, την θεωρεί ότι έχει μείζωνα σημασία και ιδίως μέσα στα πλαίσια των κινδύνων που αντιμετωπίζουμε τελευταία για την πολυφορία στην ενημέρωση. Και βλέπει ότι το περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης είναι όλο και πιο διαδικτυωμένο. Απευθύνει έκκληση λοιπόν και στο ευρωπαϊκό και στο εθνικό επίπεδο για να εξευρεθούν λύσεις στις σημαντικές, στους σημαντικούς αυτούς κινδύνους της συγκέντρωσης των μέσων ενημέρωσης, την έλλειψη ανεξαρτησίας από πολιτικές και οικονομικές πιέσεις, τα fake news, κενά στην προστασία των δημοσιογράφων και των πηγών τους, κηρύγματα μίσους, απειλές διαδικτυακά και ούτω καθεξής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντοτε τάχθηκε υπέρ της πολυφωνίας στα μέσα ενημέρωσης και στον τύπο. Πρόσφατα, με ψήφισμά του, στις 24 Δεκάτου 2017, ζητεί λήψη μέτρων για την προστασία των καταγγελόντων. Συγχαίρει τον κύριο Μαλτέζε για την εργασία του, για το σημαντικό αυτό θέμα και θεωρεί ότι πρέπει να τονιστούν ορισμένες πτυχές, όπως η ανάγκη πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης από πλευράς σημειονοτήτων, επίσης από πλευράς προσώπων με αναπηρίες. Ζητεί επαρκή χρηματοδότηση των δημόσιων μέσων ενημέρωσης για να αντιμετωπίζεται η διάδοση των ψευδών ειδήσεων πανευρωπαϊκή προστασία των καταγγελόντων, αυτών που στα αγγλικά ονομάζονται whistleblowers. Ο κ. Δεγκίτσι εντάσσει τις απόψεις του αυτές σε τροπολογίες, τις οποίες θα προωθήσει για συζήτηση με, του, με τους άλλους κοιόδης εισηγητές και τον εισηγητή. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε, η κυρία Τζίμινες Μπάμπατ. Χιμένες, Χιμένες, με συγχωρείτε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μαλτέζε για την ε, εργασία του. Ε, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και η πολυφωνία είναι θέματα τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ε, ελευθερία έκφρασης και βεβαίως όπως είπε και ο ίδιος ο εισηγητής είναι δείγμα δημοκρατίας και θα πρέπει να τα προστατέψουμε από τις πολιτικές, από τις πολιτικές επιρροές. Η εσκεμμένη διάδοση ψευδών ειδήσεων έχει δημιουργήσει εν τέλει έναν υβριδικό πόλεμο ανάμεσα στην κοινή γνώμη και την Ευρωπαϊκή Ένωση εν Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρέπει οπωσδήποτε να καταβάλει ε, κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι δημοσιογράφοι μπορούν ελεύθερα και χωρίς ε, πιέσεις από οποιαδήποτε εξουσία να, να ασκούν το λειτουργήμά τους. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ε, εν τέλει την καλή, δημοκρατία, την καλή λειτουργία της δημοκρατίας ε, σε όλες τις χώρες και σε όλες τις περιφέρειες θα μπορούσα, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσα εδώ να αναφέρω και την περίπτωση της Καταλωνίας και ό,τι έχει ακουστεί και γραφτεί γι' αυτό. Ε, θα πρέπει η δημοκρατία να προχωράει μαζί με την ελευθεροτυπία ε, την ελεύθερη και την ελευθερία της ε, έκφρασης. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται η τεκμηρίωση και η διακρύβωση των πηγών έτσι ώστε να αποφευθούν τα φαινόμενα των ψευδών ειδήσεων. Γενικά μπορώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μαλτέζε για την αξιόλογη εργασία Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο σκιώδης συγητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος τώρα, κ. Ζαμίτ. Για το συγκεκριμένο θέμα, εγώ έχω οργανώσει ε, ε στο τράπεζα για τους δημοσιογράφους στη Μάλτα και για θέματα πολυφωνίας ακούστηκαν ορισμένες απόψεις, τις οποίες θα περιλάβω και εγώ στι τροπολογίε μου, το γεγονός για παράδειγμα ότι δεν είναι μονάχα η κυριαρχία των μέσων ενημέρωση από οικονομικούς φορείς, αλλά και μάλιστα σε ορισμένες καταστάσεις και δυστυχώ έχουμε πρόσφατη εμπειρία στη Μάλτα, τα μέσα ενημέρωση δέχονται σημαντικέ πιέσει και μέσω μάλιστα νόμιμων διάβλων υποτίθεται ότι θα χρησιμοποιούνταν μια ιστοσελίδα .com προσπάθησαν να κινηθούν νομικά κατά των ε, δημοσιογράφων χρησιμοποιώντας μάλιστα νομοθεσία αμερικανική. Φανταστείτε τι θα είναι το κόστος για τους δημοσιογράφους να προσπαθήσουν δηλαδή να υπερασπιστούν τις υποθέσεις αυτές στα δικαστήρια. Άλλο θέμα που πρέπει να συζητήσουμε είναι της ποινική ευθύνη, διότι από τη στιγμή που θέματα που έχουν σχέση με τα μέσα ενημέρωσης περιλαμβάνουν και ποινικέ ευθύνε και μάλιστα και ποινέ ε, καθήξεω ή πολύ βαριών χρηματικών ποινών, αυτό, ε, κατά των δημοσιογράφων δηλαδή, αυτό έχει σημαντικέ συνέπειε στη λειτουργία των μέσων ενημέρωση. Άλλα θέματα που συζητήσαμε στη στρογγυλή αυτή τράπεζα έχουν σχέση με την βελτιωμένη προστασία των συνθήκων εργασία των ανθρώπων που εργάζονται σε εκδοτικού οίκου, μεγάλα μέσα ενημέρωση, ακόμα και αυτοί που εργάζονται ω ελεύθεροι επαγγελματίε και που συχνά το έργο τους έχει πάρα πολύ αβέβαιο χαρακτήρα και βλάπτει τον, τον επαγγελματισμό τους και βεβαίως και την ανεξαρτησία τους, ανεξαρτησία δράσεως, ανεξαρτησία σκέψης και τον τρόπο με τον οποίο ασκούν το επάγγελμά του. Άλλος παράγοντας που συζητήθηκε στην Στρογγυλή Τράπεζα ήταν τη ε, μόρφωση των επαγγελματιών, του, ε, του αλφαβητισμού των μέσων ενημέρωσης. Πρέπει να προστατεύσουμε την ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, αλλά πρέπει να δημιουργηθούν και περισσότερα προγράμματα ενημέρωσης των προσώπων, του κοινού δηλαδή, για τα διάφορα μέσα ενημέρωσης. Δέστε και τι έγραψε ο Economist πριν από λίγες εβδομάδες που έγραψε ένα άρθρο για τις ψευδείς ειδήσει και βεβαίω και την κατάσταση στο διαδίκτυο που κινείται συχνά προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που ε, για την οποία αρχικώς είχε δημιουργηθεί. Προσπαθώ να καλύψω τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν στην Τραπεζα των Δημοσιογράφων στη Μάλτα. Άλλο θέμα ήταν εάν ο έντυπος τύπος χρειάζεται τώρα περισσότερη υποστήριξη. Ο έντυπος, το έντυπο μέσο ενημέρωσης δυνοπαθεί διότι έχει ανταγωνιστές απέναντί του όλα τα ε, ψηφιακά μέσα, ενώ το ε, δημοσιογραφικό χαρτί επιβαρύνεται με δασμούς και άλλες εισφορές. Και γι' αυτό αφενός η εφημερίδα και ο έντυπο τύπο γίνεται όλο και ακριβώ, από την άλλη μεριά είναι ευθυνότερο το ψηφιακό περιεχόμενο. Αυτό όμω αποτελεί κίνδυνο και απειλή για, τις, ε, για τα έντυπα μέσα ενημέρωση και πρέπει να περιληφθεί και αυτή η διάσταση. Εν τέλει, το όλο θέμα της προστασίας του επαγγελματισμού των δημοσιογράφων. Όχι μόνο μέσω, μέσω Τη εξασφάλιση ότι δεν θα υπάρχει κυριαρχία από αυτόν, ότι δεν θα παρενοχλούνται, αλλά ιδίω όταν, ε, όσον αφορά τη δημοσιογραφική έρευνα και γνωρίζουμε, ε, γνωρίζετε την πολύ ατυχή πρόσφατη εμπειρία της δηλοφονίας τη Μαλτέζας δημοσιογράφου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται προστασία. Και όταν πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα, δεν αρκεί να αντιδρούμε απλώ, πρέπει να δρούμε και προληπτικά. Δηλαδή να προστατεύσουμε του δημοσιογράφου και όχι να έλθουμε να του υποστηρίξουμε όταν θα έχουν ήδη πέσει θύμα ε, ε, αρνητικών δράσεων σε βάρο του. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπίλτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο συνάδελφός μου για το έντυπο μέσο ενημέρωσης εκτός όταν πρόκειται για εφημερίδες οι οποίες εξακολουθούν να επιδοτούνται ενώ δεν ενδιαφέρουν πλέον απολύτως κανένα. Υπάρχουν τέτοια έντυπα στη Γαλλία και αυτό κρατά εδώ και χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να ε, υποστηρίζονται εφόσον υπάρχει. Για την ε, Μαλτέζα δημοσιογράφο δεν αρκεί ε, να ληφθούν μόνο κυρώσεις κατά ορισμένων χωρών όπως η Ουγγαρία δεν, ελήφθησαν, ε, δεν ε, επευλήθησαν κυρώσεις ούτε στην Μάλτα ενώ υπήρξαν σοβαρότατα προβλήματα κατά της ελευθερίας του τύπου και μάλιστα αυτά τα προβλήματα σημαίνονται εδώ και αρκετό καιρό. Πρέπει να γίνει προσπάθεια ήδη να αντιμετωπιστεί το θέμα. Ευχαριστώ. Uh, thank you. Uh, the committee is right to Πράγματι, η πολυφωνία των μέσων μαζικής ενημέρωσης ε, αποτελεί συνιστόσα της δημοκρατίας ε, και ειδικότερα υπάρχουν προβλήματα ε, με, το, με τα έντυπα μέσα. Υπάρχουν πολύ μεγάλες εταιρείες που έχουν κυρίαρχη ε, θέση. Εγώ πάρα πολλές φορές ε, διαπίστωσα ε, στην καθημερινότητά μου όταν υπήρχε μια ιδιαίτερη... Ήταν, ήταν υπέρμαχη του Brexit πολλές έντυπες εφημερίδες. Βλέπουμε όλο και περισσότερη αδιαλαξία από τις αριστερές εφημερίδες προς τις δεξιές εφημερίδες και υπάρχει περίπτωση τελικά να μην εισακούονται όλες οι φωνές. Ε, πολλές φορές ε, υπάρχουν μάλιστα και λαϊκιστικές προσεγγίσεις από την αναπτυξιακή πολιτική μέχρι το θέμα της μετανάστευσης. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές φορές που κάποιες αριστερές εφημερίδες ζητούν από κάποια άλλη εφημερίδα να ζητήσει συγγνώμη όταν κάνει απλώς μία προώθηση για μία πώληση σε μία συγκεκριμένη σελίδα της. Εντάξει είναι πάρα πολύ ε, δύσκολο να, να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, ε, να καταπολεμήσουμε δηλαδή αυτή την κατάσταση κατά την οποία κάποιος θέλει να κλείσει μία εφημερίδα απλώ και μόνο επειδή έχει ασκήσει κριτική. Το να εκφράσει κανείς μία γνώμη ε, δεν είναι κάτι το προβληματικό. Υπάρχει μία τάση της, αριστερά, της αριστερής πολιτικής να μην ακούει την ανταγωνιστική άποψη αλλά να προσπαθεί να απονομιμοποιήσει την έκφρασή του και δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε σε κάτι τέτοιο να συμβεί. Δεν πρέπει να του περάσει. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ε, θα ήμουν ωστόσο ευγνώμων να αφήσουμε απ' έξω αυτές τις συζητήσεις περί Brexit. Δεν εντάσσονται στο έργο της παρούσας Επιτροπής. Δεν θα επιτρέψω στο μέλλον τέτοια σχόλια. διότι βεβαίως ζήτησε το λόγο πάλι η κυρία Τζούλι Γόρντ, κάτι το οποίο νομίζω δεν προωθεί εν τέλει τη συζήτηση. Η κυρία Σάιντοβα. Ευχαριστώ αγαπητέ, αγαπητή Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συναδελφό μας Μαλτέζε για το σχέδιο γνωμοδοτήσεως. Εκτιμώ ιδιαίτερα που δίνει βάρος στην πολυφωνία και ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης. Και χαίρομαι που ομιλεί επίσης για την εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση των μέσων ενημέρωσης. Και είναι σημαντικό οι άνθρωποι να μην πέφτουν στις παγίδες των ψευδών ειδήσεων και άλλων αρνητικών φαινομένων. Κάτι όμως μου φαίνεται ότι λείπει. Εγώ θα κάνω σχετική τροπολογία, εννοώ δηλαδή την έμφαση στα δημόσια μέσα ενημέρωσης. Διότι τα δημόσια μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να αποτελούν τον εγγυητή της ανεξάρτητης ενημέρωσης που προσφέρεται σε όλα, σε όλα τα πρόσωπα, σε όλους τους ανθρώπους. Οι δημόσιοι πόροι που εισπράττονται από τις εισφορές για ραδιόφωνο, τηλεόραση κλπ. πρέπει να την χάνουν διαχείρισης απολύτως ανεξάρτητης από κυβερνήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Julie Ward. Πρώτον σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ σημαντική έκθεση. Και άκουσα με ενδιαφέρον τα περί εκπαίδευσης για τη χρήση των μέσων ενημέρωσης. Κάτι που πρέπει να εξετάσουμε είναι να δούμε πώς οι εφημερίδες χρηματοδοτούν πολιτικές θέσεις και ορισμένοι από τους μεγιστάνες του τύπου προωθούν τέτοιες θέσεις. Και απαντώ στον κύριο Φλίν, διότι το DUP που είναι ε, το αντιευρωπαϊκό κόμμα στην Βόρεια Ιρλανδία του επετράπει να κάνει δωρεά στην ε, εκστρατεία Brexit για να πληρώσει διαφημίσεις. Αυτό επετράπει μόνο στη Βόρεια Ιρλανδία, δεν επιτρεπόταν στην Μεγάλη Βρετανία. Επετράπει μόνο μέσω του διάβλου αυτού και επηρέασε κόσμο στην ε, Βρετανία. Έχουμε και ποιοτική δημοσιογραφία στην Μεγάλη Βρετανία που δυστυχώ δεν εργάζεται στην Daily Mail ούτε στην Express. Άλλοι δημοσιογράφοι που ασκούν και δημοσιογραφική έρευνα εκθέτει αυτές τις σκοτεινές ροές του χρήματος και τον τρόπο με τον οποίο υπονομεύτηκε η δημοκρατία μας. Να διαβάσετε το έργο του δημοσιογράφου αυτού, είναι εξαιρετικό. Και θα βγει, θα φανεί η αλήθεια και θα δει πώς υπονομεύτηκε η δημοκρατία μας από ακροδεξιές δυνάμεις. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Μέσερ Σμιτ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω ότι η παρούσα Επιτροπή θα επιτρέψει ευρύτερη ε, ε, συζήτηση για τα θέματα για τα θέματα της δημοσιογραφίας ε, και δεν θα βάλετε του στον κύριο Φλίν δεν συμφωνώ με τις απόψεις του, αλλά νομίζω ότι μπορεί να συζητήσει τέτοια θέματα για να δώσει παραδείγματα για το πώς λειτουργεί η ελευθερία του τύπου. Γιατί αντί να συζητούμε υποθετικά, ίσως είναι δύσκολο μέσα σε αυτή την θεωρητική συζήτηση να αντιληφθούν τα νοήματα κάποιοι που είναι λιγότερο καλοί στη φιλοσοφία όπως εγώ για παράδειγμα. Η δική μου ανησυχία σχετικά με την έκθεση και μια και εκπροσωπώ την τρίτη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα αποφάσισα να λάβω και εγώ το λόγο έστω και τώρα κάθε φορά που οι πολιτικοί μιλούν για πολυφωνία των μέσων και το τι πρέπει να κάνουν οι δημοσιογράφοι στη δουλειά του κλπ καταλήγουν τελικώς να εξασφαλίζουν λιγότερη ελευθερία και περισσότερο έλεγχο. Είδαμε πρόσφατα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδίδει εγχειρίδιο για να εξηγήσουν στους δημοσιογράφους πώς πρέπει να περιγράφουν τα μεταναστευτικά ρεύματα. Αυτό είναι λάθος. Αυτό που χρειάζεται είναι να απελευθερώσουμε τελείως τα μέσα ενημέρωσης και όχι να δίνουμε κατευθυντήρες γραμμές όπως κάνετε εσείς κυρία Πρόεδρε και όχι μόνο με τα όσα λέτε αλλά και με τις εκφράσεις του προσώπου σας που βρίσκω σαγηνευτικές κατά τα άλλα. Βρίσκω λοιπόν ότι θα πρέπει με την έκθεση αυτή να περιστούμε σε αυτά που είπα διότι αυτό χρειάζεται η δημοσιογραφία στην Ευρώπη όχι μόνο αυτά που κάνουν κάποιες κυβερνήσεις όπως Πολωνία, Ουγγαρία κλπ. Αλλά να απελευθερωθούν και από, οποιασδήποτε, από δεσμά και επιρροή από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Έτσι πρέπει να εξασφαλιστεί η ελευθερία του τύπου στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας κοίταξα λίγο παράξενα γιατί εξεπλάγιν που είπατε ότι η Κομισιόν έχει εκδώσει εγχειρίδιο που Προδιαγράφει στους δημοσιογράφου πώ θα λειτουργούν. Ο καλός δημοσιογράφος ξέρει τι θα πρέπει να κάνει. Δηλαδή, απολύτως απλά να το αγνοήσει τον κύριο Η Σίλβια Κώστα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συναδέλφο ε, Μαλτέζα για την εξαιρετική βάση ε, που έχει ε, ξεκινήσει για αυτό το πολύ θεμελιώδες, σημαντικότατο θέμα της ε, ε, πολυφωνίας και της ανεξαρτησίας. Νομίζω ότι μπορώ να συμμεριστώ τις απόψεις του και τις κρίσεις του. Νομίζω ότι εδώ ε, αυτό το κείμενο μπορεί να αποτελέσει και μία έκκληση έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε να προωθηθούν δηλαδή θέλω να πω οι απαραίτητες προϋποθέσεις ισοτιμίας διαφάνειας διαφάνειας και σαφήνειας. Ε, γιατί διαφορετικά, όπως πολλές φορές και επανειλημμένα έχω πει, ε, ε, κινδυνεύουμε στην ψηφιακή ε, Ευρώπη να δημιουργήσουμε κάποιες λεωφόρους ας πούμε της μετακίνησης της διάδοσης της πληροφορίας αλλά να μην έχουμε όλοι τις ίδιες ευθύνες. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά το, περιεχόμενο, όχι φυσικά εν είδη λογοκρισίας. Πιστεύω ότι η ο αντίκτυπος ε, της ελλειπούς ε, πολυφωνίας που την ε, διαπιστώνουμε ε, με, την, ε, με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι εκδότες, η εκδοτική οίκη που αποτέλεσε πλούτο της Ευρώπης και με την διάδοση αυτών των ψευδών ειδήσεων όχι μόνο και λόγω της έκκλησης που πρέπει να γίνει προς όσον αφορά τις πολιτικές δυνάμεις αλλά και λόγω των πολλών αντικτύπων που μπορεί να έχει, όπως έλεγε και η Στέλφος, Χιμένες. Ε, νομίζω ότι πρέπει να θυμίσουμε ας πούμε, ότι στην ε, ε, χώρα μου συχνά έχει γίνει λόγος και για μια επιστημονική αρχή, scientific authority, η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει ενδεχομένως. Ε, τι να σας πω τώρα, υπάρχουν ε, ψευδείς ειδήσει ακόμα και για θέματα καθαρά επιστημονικά, όπως ας πούμε ε, μέσα από διάφορες εκστρατείες μέσω του τύπου και απόψεις που εκφράζονται μέσω του τύπου, έχει μειωθεί κατά 30% ο εμβολιασμό των παιδιών, ας πούμε, το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει και συνεργασία με γειτονικέ χώρες και συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών, αλλά και χώρες Όπω συνέβη πρόσφατα και με τα Τύρανα, με συνεργασία με χώρες γειτονικέ, με χώρες ε, που έγκυται στι ε, πολιτικέ γειτονίε κτλ. Ε, και τέλος, όσον αφορά τις δημόσιες, τους δημόσιους διάβλους, θα πρέπει να διατηρηθούν, είναι πάρα πολύ σημαντικοί, μπορούν να αποτελέσουν εχέγγυο αντικειμενικότητας αλλά και βοήθεια και για τι τοπικέ τηλεοράσει. Πιστεύω ότι θα μπορούν να γίνουν και κάποιε αναφορέ όσον αφορά ε, την ελεύθερη πρόσβαση στην ε, πληροφορία μέσα από μεγαλύτερη συνεργασία όλων των εργαζόμενων και του κλάδου. Ευχαριστώ πολύ. Bardzo dziękuję. Padało tu parokrotnie zdanie, że media są filarem demokracji. Tak, są filarem... Ευχαριστώ αγαπητή Πρόεδρε. Θα πρέπει, όπως είπαν και άλλοι, η δημοσιογραφία να είναι απολύτως ανεξάρτητη και ελεύθερη, γιατί αλλιώς γίνεται όργανο χειραγώγησης. Συμφωνώ με την κυρία Σόντροβα. Τα δημόσια μέσα ενημέρωσης πρέπει να είναι απολύτως πολύφωνα. Γιατί η δική τους ευθύνη είναι να φροντίζουν η αποστολή τους να είναι ευρύτατη και η πολιτική και η κοινωνική. Αυτό οφείλουμε να το απαιτήσουμε. Δεύτερο, οι δημοσιογράφοι. Θα συμφωνήσω με την κυρία Χιμένες ότι οι δημοσιογράφοι όλο και περισσότερο βρίσκονται σε κίνδυνο. Υπάρχει μια τέτοια τάση. Εξάλλου η εργασία τους είναι αβέβαιη. Οι συμβάσεις εργασίας με τις οποίες εργάζονται είναι αβεβές. Δεν υπάρχει λογοκρισία βέβαια στην Ευρώπη, υπάρχει όμως η λογοκρισία που επιβάλλει ο εκδότης. Εν τέλει, τα ψηφιακά μέσα. Εδώ υπάρχει ένα είδος χάσμα των γενεών. ο έντυπος τύπος, η, έντυ, έντυπη εφημερίδα διαβάζεται κυρίως από τη μεγαλύτερη γενιά. Τα ψηφιακά μέσα από τους νέους. Όμως, τελικώς θύματα πέφτουν της χειραγώγησης κυρίως οι πιο ηλικιωμένοι, διότι δεν έχουν τη δυνατότητα ή δεν έχουν τη γνώση να ψάξουν μέσα στο διαδίκτυο να βρουν και άλλες απόψεις. Πρέπει να δοθεί τέλο να γίνει προσπάθεια και για την εκπαίδευση των ίδιων των δημοσιογράφων. Ο κύριο Διακόνου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λέχθηκαν πολλά έω τώρα. Έχουμε την έκθεση του κυρίου Μαλτέζη που θεωρώ ότι είναι καλή και θα αποτελέσει επιτυχία. Διακόνου κόπτει μια άλλη συνάδελφος από κάτω χωρίς μικρόφωνο και δεν την ακούμε ό,τι αυτήν ούτε τον κύριο Διακόνου. Ο κύριος Διακόνου πάλι. Ευχαριστώ. Θα πω μόνο ένα πράγμα. Απευθύνοντάς σας μια πρόκληση και εκφράζοντας μια ανησυχία. Κάθε ήχος που ακούγεται στη φύση έχει και την ηχό, μια αντίχηση. τα, τα μέσα ενημέρωσης παράγουν και αυτά ήχους. Και αυτοί είχε έχουν πάλι αντίχηση. Που είναι σημαντική, το εννοώ μεταφορικά βέβαια. Όταν μιλούμε για τα νέα, για τις ειδήσει, η αντίχηση είναι διαφορετική. Εξαρτάται από την υπευθυνότητα, η αντίχηση αυτή, των μέσων που καμιά φορά προσπαθούν να προκαλέσουν διαφορετική αντίχηση. Και είναι δύσκολο να κατανοήσουμε πού βρίσκεται το όριο ανάμεσα στα υπεύθυνα μέσα ενημέρωσης και στην αντίχηση με αυτή που έρχεται μέσα από το σκοτάδι, μέσα από blog, από bloggers και ούτω Αυτό το σκοτάδι είναι που τροφοδοτεί τις ψευδείς ειδήσει. Προσπαθούν να αλλάξουν την πραγματικότητα. Εδώ βρίσκεται νομίζω η πραγματική πρόκληση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη Σαμπίνε, ε, παρανόηση υπήρξε. Είδα την κυρία Σόιντροβα πριν, τώρα σε είδα εσένα και κάπου δεν κατάλαβα ότι ζήτωσες το λόγο. Τι χαίρομαι πολύ που μας συγχαίει στην κυρία Σόιντροβα και εμένα, αλλά μιας και μιλήσαμε για πολυφωνία, να ακουστεί και η δική μου φωνή. Και πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο Μαλτέζε για την έκθεσή του. Γνωρίζω ότι βεβαίως ε, υπάρχει περιορισμό των σελίδων στην έκθεση γνωμοδότησης και υπάρχει πίεση να περιληφθούν πολλά πράγματα. Και αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι με τις μεγάλες αλλαγές στην ψηφιοποίηση των μέσων αντιμετωπίζονται και σημαντικές προκλήσεις και για τους δημοσιογράφους, διότι η διαφορά πλέον ανάμεσα στα καθιερωμένα ποιοτικά φύλλα και την ποιοτική δημοσιογραφία και κάποιον οποιονδήποτε ο οποίο εμφανίζεται και δηλώνει δημοσιογράφο και γράφει κάτι στο διαδίκτυο. Λοιπόν, η διάκριση αυτή είναι δύσκολο να γίνει. Δηλαδή πολλοί εμφανίζονται στο διαδίκτυο με ειδήσει χωρίς να διαθέτουν ούτε το ποιόν, ούτε την ε, εκπαίδευση του δημοσιογράφου και γι' αυτό συμφωνώ με την κυρία Λιμπάτσκα. Χρειαζόμαστε εκπαίδευση του τύπου, των δημοσιογράφων, των μέσων, αλλά χρειαζόμαστε και θαραλέους δημοσιογράφους. Η δημοσιογραφία ήταν κάποτε ένα επάγγελμα το οποίο πληρωνόταν καλά, το οποίο ε, δημιουργούσε πραγματικά έργο ουσίας με καλά εκπαιδευμένους δημοσιογράφους. Σήμερα πολλοί δημοσιογράφοι είναι υποχρεωμένοι να είναι αναγκασμένοι να, να αρκεστούν στο απόλυτο ελάχιστο. Δεν σημαίνει ότι όποιο δημοσιογράφος πληρώνεται άσχημα είναι και κακό δημοσιογράφος. Το τονίζω και το υπογραμμίζω αυτό. Αλλά παίζει κάποιο ρόλο. κάποιο ο οποίο πρέπει να αποδώσει καλό έργο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα και οικονομικά επομένως να έχει εξασφαλισμένο το προστοζήν ώστε να μπορεί να κάνει και την έρευνα. Αυτό, αυτή η υποχρέωση βαρύνει τους επιχειρηματίες του τύπου. Πρέπει να θεσπίσουν τις αναγκαίες συνθήκες πλαίσια ώστε να μπορούν οι δημοσιογράφοι να εργαστούν οικονομικά ανεξάρτητοι. Θεωρώ λοιπόν ότι το ζήτημα αυτό είναι σημαντικό. Ταυτόχρονα σημαντική είναι και η ιδεοντολογία του δημοσιογράφου. Ποια είναι η ευθύνη του τέταρτου πυλώνα εξουσίας ή τέταρτης εξουσίας αν θέλετε. Δεν μπορώ να πιάνω οποιαδήποτε ιστορία μου έρθει στα αυτιά να την αναμεταδώσω ακρίτως. Χρειάζεται να γίνει αξιολόγηση της είδηση και χρειάζεται κυρίως να γίνει διασταύρωση και διερεύνηση της είδηση. να απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις ο δημοσιογράφος πρώτα, στο απέναντι στον εαυτό του δηλαδή, πριν προχωρήσει η δημοσίευση της είδηση. Και νομίζω ότι εδώ τα μέσα έχουν τεράστια εξουσία, η τάση που διαγράφεται είναι και μεγάλη πίεση προς την δημοσιογραφία, τα βλέπουμε αυτά και στην Πολωνία και στην Ουγγαρία, όπου οι ασκούντες στην εξουσία ανησυχούν ότι κινδυνεύουν από τη δράση των μέσων και το πρώτο τους βήμα είναι να τα υποτάξουν. Αυτό καμιά φορά γίνεται μέσω οικονομικών πιέσεων δεν εξηρώ την Μάλτα και νομίζω ότι θα πρέπει να πω στους ε, Μαλτέζους φίλους μου ότι το Κοινοβούλιο το ίδιο, το Ευρωπαϊκό δηλαδή, έχει ψηφίσει ψήφισμα για την Μάλτα. Δεν κλείνουμε δηλαδή τα μάτια απέναντι στην πραγματικότητα αυτή. Ο πολίτης έχει δικαίωμα ενημέρωσης και απέναντι σε αυτό το δικαίωμα αντιστοιχεί η υποχρέωση του δημοσιογράφου που χρειάζεται όμως εξασφάλιση ποιότητας, πολυφωνίας και πρέπει εμεί εν τέλει νομοθετικά να φροντίσουμε να υπάρξουν τα αναγκαία πλαίσια στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρο Κάμερ Εβερτ. Βρήκα τη συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα. Τόνισε τι διαφορετικέ πτυχέ που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ανεξαρτησία των μέσων, εκπαίδευση των δημοσιογράφων, ποια είναι η οικονομική κατάσταση των δημοσιογράφων αλλά και των εφημερίδων, ανεξαρτησία των μέσων, πολυφωνία των μέσων, όλα αυτά παίζουν στο πλαίσιο αυτό πολύ σημαντικό ρόλο. Επισημαίνω μόνο ότι στην έκθεση μπορούμε να γράψουμε όλα όσα συζητήθηκαν εδώ, αλλά αποκλειστική αρμοδιότητα έχουμε μονάχα για περιορισμένη. Δηλαδή αν μιλήσουμε για ανεξαρτησία των μέσων, η ελευθερία των μέσων, Μπορούμε να τα κάνουμε, δεν μπορούμε να απαιτήσουμε όμως από την Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών να τα περιλάβει αυτούσια όσα τα πούμε στη γνωμοδότησή μας. Ό,τι πούμε για τα μέσα, διακόπτη η συνάδελφος από ε, κάτω χωρίς ε, μικρόφωνο, εμείς ως Επιτροπή έχουμε αποκλειστικά αρμοδιότητα μόνο για την αρμοδιότητα των μέσων. Δεν έχουμε για πολυφωνία και ελευθερία. Εκεί την αρμοδιότητα έχει η Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών. Άρα, ξαναλέω, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, αλλά η αρμοδιότητά μας εξαντλείται να μιλήσουμε μονάχα για την, ό,τι, έχει, ό,τι είναι αρμοδιότητα των ίδιων των μέσων. Για παράδειγμα, εκπαίδευση δημοσιογράφων. Το υποδεικνύω αυτό, ότι χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στο ποιο είναι το περιεχόμενο μιας απλής γνωμοδότησής μας και ποια είναι η δική μας αρμοδιότητα. Τώρα, κανονικά θα έπρεπε να έχουμε και εκπρόσωπο της Κομισιόν, επειδή όμως το προτάξαμε το θέμα αυτό, α, η κυρία Σαμπίνε Φερχάιν, δεν είναι πιο απλό να χωρίσουμε τη γνωμοδότηση σε δύο κεφάλαια και στο ένα κεφάλαιο να αναφερθούμε μοναχά σε αυτά όπου έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα και μετά στο υπόλοιπο της νομοδοτήσεως να υποβάλουμε κάποιες σκέψεις μας στην Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών. Να μην έρθει δηλαδή η Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών και διαγράψει όλα όσα γράφουμε τελικώς στη γνωμοδότησή μας. Ένα τμήμα λοιπόν μονάχα για όσα έχουν αποκλειστικά σχέση με τα μέσα την, την ικανότητα δηλαδή των μέσων να εκπαιδεύουν δημοσιογράφου κλπ. Και τα υπόλοιπα να τα βάλουμε ξεχωριστά. Μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό θα είναι βέβαια το καθήκον του εισηγητού και των σκιωδών εισηγητών να χωρίσουν τα πράγματα έτσι ώστε να είναι σαφώς αναγνωρίσιμα που θεωρούμε ότι τα θέματα άπτονται της δικής μας αποκλειστικής αρμοδιότητας και που απλώς υποβάλλουμε γνωμοδότηση στην Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών με την παράκληση να το λάβει υπόψη της. Είμαι βεβαία ότι πολλά από τα όσα συζητήσαμε θα συζητηθούν με τον ίδιο περίπου τρόπο και, τρόπο και στην Επιτροπή Θεμελιδών Ελευθεριών. Θα χαρούν λοιπόν τα μέλη της Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθεριών να ακούσουν και δικές μας προτάσεις. Αλλά, όντως, να γίνει ο διαχωρισμός των αποκλειστικών μας αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 53, αλλά αυτά μπορούν να γίνουν στα πλαίσια της τεχνικής διαδικασίας και στις διαβουλεύσεις ή διαπραγματεύσεις για τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Θα δώσω το λόγο πάλι σύντομα. Βλέπω πάλι εκεί από, στα έδρανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να λάβει το λόγο για το θέμα αυτό. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώ ε, το βάλαμε πιο μπροστά το θέμα αυτό. Δεν απευθύνω απολύτως καμία μομφή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχεις και πάλι το λόγο αγαπητέ Κούρτσιο. Ε, Ευχαριστώ. εξ όσων γνωρίζω και από τους συναδέλφους της ΛΥΜΠΕ δεν νομίζω ότι θα ζητήσουν ε, άσκηση ε, αποκλειστικής αρμοδιότητας όσον αφορά την πολυφωνία. Είναι μάλλον πλουραλιστές και πολυφωνικοί όσον αφορά το θέμα αυτό. Ε, το ζήτημα το οποίο έδειξαν περισσότερο οι συνάδελφοι είναι αυτό της κατάρτισης, της εκπαίδευσης στα μέσα ε, ενημέρωσης. Αυτό και ορθώς έχουν επικεντρωθεί σε αυτό. Η ιστορία της πληροφόρησης και της πληροφορίας ε, είναι πραγματικά γεμάτο από τέτοιες μικρές επαναστάσεις και στην αρχή ας πούμε λέγαμε ότι το ραδιόφωνο θα σκότωνε κατά κάποιο τρόπο τον γραπτό τύπο ή ότι η τηλεόραση μετά με τη σειρά της θα δολοφονούσε το ραδιόφωνο κτλ. Αλλά ε, είδαμε ότι ε, στην ουσία σιγά σιγά ε, το κοινό εκπαιδεύτηκε στη χρήση των νέων μέσων. Τώρα έχουμε νέα μέσα ενημέρωσης, τα οποία όμως έχουν διαχύσει την ε, ιδέα ότι ε, είναι πιο εύκολο να ε, πληροφορείται κανείς μέσα από τα πιο εύκολα κανάλια, μέσα από διάβλους που είναι πολύ πιο ε, απλοί κτλ. Τώρα, όνο, όμως αναδύονται τα fake news, οι ψευδείς ειδήσει. Όταν εγώ χρησιμοποιώ ας πούμε την Wikipedia για να, να ψάξω κάτι το οποίο όμως το γνωρίζω καλά διαπιστώνω ότι υπάρχουν πάρα πολλές εσφαλμένες πληροφορίες και όμως ε, ε, ε, πλανητικά είναι η πηγή, η Wikipedia, την οποία, από την οποία ενημερώνεται ο περισσότερος κόσμος. Πρέπει να διαπιστώσουμε αυτό το στοιχείο και θα πρέπει οπωσδήποτε να το αναφέρουμε γιατί είναι κάτι το οποίο αποτελεί πρώτη και κυρίαρχη δική μας αρμοδιότητα να το κάνουμε αυτό. Βεβαίω, και για του επαγγελματίε δημοσιογράφους αλλά και για όλους είναι δύσκολο να ε, βρουν και να απομονώσουν αυτά τα εργαλεία τα οποία θα επιτρέψουν την εκπαίδευση του κοινού ε, στα νέα μέσα ενημέρωσης. Ευχαριστώ. Η ε, Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι στους σκιώδεις και στον εισηγητή καλή δουλειά, πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και μια καλή γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ. Με το θέμα αυτό τώρα λοιπόν ολοκληρώσαμε. Έχουμε το πρόβλημα τώρα ότι δεν είναι παρόντες οι βραβευθέντες, γι' αυτό θα αναγκαστώ να διακόψω σύντομα. Σας παρακαλώ όμως μείνετε εδώ ή πάντως κάπου κοντά στην αίθουσα. Διότι έχουμε δει στο παρελθόν να είναι κάπως άδεια η αίθουσα όταν πρόκειται για την ε, απονομή ή τέλος πάντων για την συζήτηση με τους βραβευθέντες του Καρ Χάιντς Θα ήθελα να σας παρακαλέσω λοιπόν να είστε εδώ. Θα διακόψω την συνεδρίαση αλλά μην απομακρυνθείτε. Christina, bitte. Ε, Κριστίνα. Ευχαριστώ. Πότε αναμένετε τους βραβευθέντες. Εγώ θέλω να είμαι παρούσα. Αλλά 11 η ώρα έχω άλλη συνάντηση. Στις 10 είχαν συνάντηση με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Ταγιάννη για την ε, παραδοσιακή φωτογραφία. Καμιά φορά αυτό μπορεί να κρατήσει λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά νομίζω σε Πέντε το πολύ 10 λεπτά θα είναι εδώ τα πρόσωπα αυτά. Άρα λοιπόν κινηθείτε αναλόγως. Διακοπή πέντε λεπτών.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

θα ήθελα να σας ζητήσω να σταματήσετε τις συζητήσεις σας ή αν θέλετε να τις συνεχίσετε, απλώς να αποχωρήσετε από την αίθουσα. Είναι πολύ μεγάλη χαρά να συνεχίζουμε την ε, παράδοση που έχουμε κάθε χρόνο. Υποδεχόμαστε τους ε, βραβευθέντες, τους νικητές του βραβείου Καρλομάγνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέτος θα βγούμε από τη συνηθισμένη μας διαδικασία γιατί είναι η δέκατη επέτειος του βραβείου αυτού οπότε σήμερα είναι εδώ ε, οι νικητές του βραβείου από το 2008. Καλώς ήρθατε. Όλοι οι νικητές ε, έχουν ήδη παραστεί για την ε, απονομή του βραβείου τους και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είναι παρόντες και πάλι σήμερα. Χωρίς ε, να καθυστερήσω άλλο, θα, σας θα δώσω τους το λόγο στους νέους που έλαβαν τους, το βραβείο σήμερα, φέτος, του 2017. Πολωνία, Δανία και κάτω χώρες είναι οι νικητές. Erasmus Evening από την Πολωνία είναι το, πρόγραμμα, το, ε, το πρόγραμμα που νίκησε φέτος. Θα δώσω το λόγο ε, στους νέους για να το παρουσιάσουν. Είναι ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα, ένα ε, μέσο το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Σκοπό έχει να ενημερώνει ε, τους νέους για την δυνατότητα σπουδών στο εξωτερικό και να τους ενημερώνει επίσης και για τις καλές εμπειρίες του Εράσμους. Ο στόχος είναι να προσπαθήσουμε να ενημερώνουμε περισσότερο τους νέους. Ο τελικός στόχος είναι να προωθήσουμε την αμοιβαία κατανόηση, τον διαπολιτισμικό διάλογο και να ε, ξεπεράσουμε ε, τα ε, πνευματικά εμπόδια. Τρίτος, τρίτο βραβείο, Rediscovering Europe, Μόνικα Έλεντ από τις κάτω χώρες. Σκοπό έχει να υποστηρίξει τις δεσμεύσεις ε, των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε μια περιοχή της Δανίας μέσω δράσεων, συζητήσεων, ε, παρελάσεων, εορταστικών εκδηλώσεων. Πάνω από τέσσερις ε, πάνω από 40 εθελοντές συγγνώμη, συμμετείχαν στην όλη διαδικασία για να μπορέσουν να ενισχύσουν ε, το φιλοευρωπαϊκό αίσθημα των ε, πολύ ευροσκεπτικιστικών περιοχών. Η Γκίς Κισελ από την Ολλανδία. Και τα πρόσωπα αυτά έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν απόψεις, να κινητοποιήσουν νέα πρόσωπα να αναπτύξουν ένα νέο θετικό αφήγημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το πώς σκέπτονται οι νέοι περί Ευρώπης και πώς ταυτίζονται όσο ταυτίζονται μαζί της. Εν τέλει, έχουμε λίγο λιγότερο από μια ώρα για την παρουσίαση των σχεδίων. Γι' αυτό, χωρίς περισσότερα λόγια, να δώσω το λόγο αμέσως στους νεαρούς προσκεκλημένους μας και στις νεαρές προσκεκλημένες Νομίζω εν τέλει κερδισμένοι είναι όλοι και κυρίως η Ευρώπη από αυτή την πραγματικά θαυμάσια δέσμευση νέων ανθρώπων υπέρ του ευρωπαϊκού εγχείρηματο. Και πρώτα βέβαια, ή μάλλον ε, τα τελευταία μου λόγια είναι τα συγχαρητήρια, θερμότατα συγχαρητήρια στους νέους και στις νέες που έχουμε κοντά μας. Αρχίζουμε με την παρουσίαση του σχεδίου Erasmus Evening από την Πολωνία, η κυρία Γέλονεκ για 7 λεπτά. Στα αγγλικά. Θα προσπαθήσω να σα τα πω στα αγγλικά. Το, η ραδιοφωνική μου εκπομπή ήταν επίση στα αγγλικά. Έχω και μία παρουσίαση, αλλά άραγε θα λειτουργήσει. Θα έπρεπε να αρχίσει τώρα. Η ανάγκη μας κάνει εφευρετικούς. Εγώ υπήρξα δύο φορές σπουδάστρια έρασμος. Πρώτη φορά το 2014 με το πρόγραμμα LOP. Μετά έγινε έρασμος ΣΥΝ. Είχα λοιπόν κάποιες εντυπώσεις κομίση για το πώς λειτουργεί το πρόγραμμα και ποιες είναι οι αλλαγές, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα κάποιες φορές και ήθελα να δημιουργήσω ας πούμε ένα χώρο όπου οι άνθρωποι να μπορούν να εκφράσουν όποια άποψη επιθυμούν, ε, να παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους. Και αντιλήφθηκα ότι εάν επιθυμεί κανείς να αναζητήσει πρακτικές προφορίες για το πρόγραμμα Έρασμος, πρέπει να πάτε στο διαδίκτυο, blogs, πλατφόρμες και να καταναλώσετε πολύ χρόνο στη σχετική έρευνα εγώ εργαζόμουν στο ραδιοφωνικό σταθμό των φοιτητών, Radio Meteor, όπως βλέπετε στην ε, διαφάνεια που τώρα δεν λειτουργεί δυστυχώς, δεν, δεν ε, προβάλλεται. Καλά, ίσως αργότερα. Έτσι λοιπόν Και καμιά φορά δυστυχώ έχουμε διακοπέσει το μικρόφωνο τη ομιλήτρια. Δεν ακούμε. Τώρα την ακούμε πάλι. Και για να αντιμετωπίσετε τα διάφορα προβλήματα που δεν είναι πάντοτε εύκολο να ρυθμιστούν. Για παράδειγμα, στη δική μου περίπτωση πήγα στην Ισπανία μετά το πανεπιστήμιο μου είπε «Α, δεν έχουμε τα χαρτιά σας» και άρα δεν είστε φοιτητή έρασμο. Χρειάστηκε να περάσει, περάσουν κάποιες εβδομάδες μέχρι να έρθουν τα χαρτιά μου. Κάποια στιγμή ε, συμβαίνουν τέτοια πράγματα και εδώ έχω ε, ε, πρόσωπα από τη Γεωργία και την Ιταλία στη φωτογραφία. Η κοπέλα που βλέπετε είναι από το Καζακστάν. Μιλούμε και για τα έθιμα, για την καθημερινή ζωή, διότι όταν πάτε κάπου αρχίζετε, να είστε μέρο, μέλος μιας κοινότητας. Και μιλήσαμε και για το κοινωνικό πρόγραμμα Erasmus, ε, διότι το βασικό είναι όταν πάτε κάπου δεν είναι τόσο οι σπουδές η, η ανακάλυψη μιας νέας χώρας ή νέας πόλης μπορείτε να αφήσετε και τη σφραγίδα σας μπορείτε να βοηθήσετε ανθρώπους να μάθουν ξένες γλώσσες για παράδειγμα στην Πορτογαλία στο δεύτερο έρασμος που συμμετείχα Ορισμένοι δίδασκαν την κιθάρα ή ξένες γλώσσες. Μπορείτε λοιπόν να μοιραστείτε με τους άλλους αυτό που διαθέτετε και κυρίως το χρόνο σας μια φορά το πιο σημαντικό. Πήγαμε και μαζεύαμε φίλια με ηλικιωμένους για να τους βοηθήσουμε να ε, φτιάξουν διάφορα πράγματα ή ε, αγοράζαμε υγιεινά προϊόντα για να τα δώσουμε σε ηλικιωμένους. Όταν πάτε κάπου μπορείτε να μοιραστείτε μαζί τους ό,τι θέλετε, ό,τι διαθέτετε και αυτό σημαίνει ότι είμαστε διαφορετικοί από εσά, αλλά όλες οι χώρες, όλες οι εθνικότητες έχουν κάποια κοινά πράγματα. Και αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι να δείξουμε στους ανθρώπους ότι μπορούμε εύκολα να πάμε να ενταχθούμε σε μια κοινότητα και να επανέλθουμε ευφιέστεροι με λιγότερες προκαταλήψεις, με λιγότερα στερεότυπα, γιατί αν δεν έρχεστε σε επαφή με άλλους ανθρώπους, αν δεν συνεργαστείτε με άλλους ανθρώπους, μάλλον είναι δύσκολο να τους κατανοήσετε και να δουλέψετε μαζί τους. Και από τη δική μου δουλειά, άνθρωποι που δεν πάνε στο εξωτερικό και είναι πάντοτε, ζουν πάντοτε στην ίδια πόλη, δεν ανοίγει το μυαλό τους. Όταν έχουν μια ιδέα, την κρατούν για τον εαυτό τους και δεν ακούν και τι λένε οι άλλοι. Όταν μπείτε στο Εράσμος όμως, αναγκάζεστε να συνεργαστείτε με τους άλλους ανθρώπους. Κατά τη γνώμη μου, ο Εράσμος θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικός για όλους και όλους. Και στο, στην εκπομπή μας δείχνουμε ότι αυτό το πρόγραμμα βοηθεί να ανοίξει το μυαλό των ανθρώπων. Βλέπετε να ορισμένοι ήρθαν και τραγουδήσανε στην ραδιοφωνική μας εμπειρία και αγρότες. Έχουμε και προφίλ στο facebook, Erasmus Evening λεγόμαστε, γιατί ορισμένοι προσπαθούν, κάποια άτομα δηλαδή στο διαδίκτυο προσπαθούν να φτιάξουν ένα ψεύτικο προφίλ, παίρνοντα και δικά σας στοιχεία. Έχουμε εδώ και ε, τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν θέλετε μπορείτε να παρακολουθήσετε γιατί τα βγάζουμε και στο YouTube αυτά. Έχω και ένα blog όπου βάζω πληροφορίες για το έρασμος και νέες ειδήσει. Και αυτά, αυτή είναι η τελευταία διαφάνεια. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πέτρα Κάμερ Εύερτ Βλέπω ότι επενείτε πολύ τον έρασμο και είστε πολύ ενθουσιώδεις. Νομίζω να την κάνουμε πρέσβη υπέρ του έρασμους για να πείσουμε και το Συμβούλιο Υπουργών ότι χρειαζόμαστε περισσότερη χρηματοδότηση για το έρασμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ήλεντ με το project ανακαλύπτουμε την Ευρώπη από τη Δανία. Επτά λεπτά για να παρουσιάσετε το πρόγραμμα σας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχά να πω ότι χαίρομαι όλο ιδιαίτερος που εκπροσωπώ αυτό το ε, πρόγραμμα τη Δανία που πήρε τη δεύτερη θέση στο βραβείο Κάρλο Μάγνου. Ε, είμαι ε, Πολωνή αλλά ζω στην Δανία εδώ και έξι χρόνια και γι' αυτό έχω ένα πολύ ευρωπαϊκό αίσθημα. Το πρόγραμμα η νέα ανακάλυψη, ξανανακαλύπτουμε την Ευρώπη, προέκυψε επειδή θεωρήσαμε ότι υπάρχει μια ανάγκη να επενθυμίσουμε στον κόσμο τι θα πει ενωμένη στην πολυμορφία ε, Είναι μια πόλη, το Ότμπουργκ, στη Βόρεια Δανία. Το 2016 ε, βαθμολογήθηκε ως η πιο ευτυχισμένη πόλη στην Ευρώπη. Είναι, είναι επίσης μια πόλη που, στην οποία ζουν πάνω από από 50 εθνικότητες και θέλουμε να δείξουμε ακριβώς ε, πόσο σημαντικό είναι το να ζει κανείς σε μια κοινωνία. Η Ευρώπη χρειάζεται τέτοιου είδους ιστορίες, επιτυχημένες ιστορίες ε, <clears throat> σωστής ενσωμάτωσης και ένταξης. Ε, καταρχάς προσπαθήσαμε να οργανίσουμε μια πολιτιστική παρέλαση, Pride of Cultures, ε, ενωμένη στην πολυμορφία. Υπήρχε φαγητό, μουσική, ε, χωρί. Καλέσαμε όλες τις πολιτιστικές ομάδες, τους διαφόρους συλλόγου, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, πάνω από 16 διαφορετικές ομάδες. Δεν είναι πάρα πολλέ από τις 155, αλλά ε, το επαναλάβαμε και φέτο και φέτο τα πήγαμε πολύ καλύτερα. Δεύτερο τμήμα του προγράμματός μας ε, ήταν ε, η εστίαση στην ενημέρωση. Οργανώσαμε μία σειρά δραστηριοτήτων την ημέρα τη Ευρώπη, ώστε να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Μιλήσαμε με κόσμο στο δρόμο, δώσαμε υλικό, ε, είχαν κάποιοι μάλιστα μεταμφιεστεί, κάναμε πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε την προσοχή και αυτό ακριβώς, ε, σε αυτό ακριβώς συνίσταται το, πρόβλημά μας, το πρόγραμμά μας να ενημερώσουμε την Ευρώ, τον κόσμο για την Ευρώπη και να έχει μια εμπειρία της Ευρώπης. Προσπαθήσαμε λοιπόν με την ευκαιρία αυτή να δείξουμε τι μας δίνει αυτό το πρόγραμμα. Μας ενέπνευσε να κάνουμε πολύ περισσότερα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να ε, αισθάνεται ο κόσμος ότι συνδέεται πιο πολύ, ε, έχει μια σχέση με την κοινωνία. Ε, να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να μετακινείται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Αυτό που θα ήθελα επίσης να πω ότι τον τελευταίο 1,5 μήνα υπήρχαν τοπικές και περιφερειακές εκλογές στην Δανία και παρά το γεγονός ε, ότι η προσέλευση είναι συνήθως υψηλή, ρωτήσαμε τον κόσμο ε, τι γίνεται με τους μη δανούς, ε, πώς γνωρίζουν ότι έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν και εκείνοι. Ε, ήρθαμε λοιπόν σε επαφή, στοχεύσαμε κυρίως τους φοιτητές. Πολύ λίγοι γνωρίζουν ότι έχουν το δικαίωμα ψήφου. Αυτό διαπιστώσαμε παρά το γεγονός ότι ζουν εκεί τόσα πολλά χρόνια. Πολλοί κόσμος ε, έρχεται για σπουδές αλλά παρόλα αυτά μετά στη συνέχεια παραμένει για δουλειά, έρχεται η οικογένειά του αλλά θεωρούν ότι επειδή δεν είναι δανεί δεν μπορούν να ψηφίσουν. Και όμως μπορούν να ψηφίσουν. Οπότε οργανώσαμε μία εκστρατεία στα αγγλικά ε, υπήρξε υλικό, έντυπα, ε, τυπώσαμε τα δικαιώματά τους, τους εξηγήσαμε ότι ε, μπορούν και για ποιο λόγο πρέπει να ψηφίσουν. Και πρέπει να πω οι εκλογές τελείωσαν εχθές. Χθες ε, ήταν η μέρα της ε, ψηφοφορίας. Ε, τελείωσε η προεκλογική εκστρατεία και ελπίζουμε ότι θα φανεί η προσπάθειά μας και στα αποτελέσματα. Ελπίζουμε ότι η προσέλευση θα είναι πολύ ψηλότερη μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών, ε, γιατί ε, το θέμα είναι δεν, ότι δεν πηγαίνει κανεί σε μία άλλη χώρα για να δουλεύει, να είναι τμήμα, να έχει μία κοινωνική ζωή, αλλά πρέπει να συμμετέχει και στον πολιτικό βίο. Είναι πολύ σημαντικό τρόπο να μπορεί κανείς και να συνεισφέρει και να δείχνει ε, ότι συμμετέχει σε αυτή τη νέα κοινότητα στην οποία έχει επιλέξει να ζήσει. Αυτό κάναμε μας ενέπνευσε να κάνουμε ακόμη περισσότερα και ελπίζουμε ότι θα ε, φέρει την αλλαγή Υπήρξε κάποια προσοχή μάλιστα και από τα εθνικά μέσα της Δανίας, ε, μέσα ενημέρωσης της Δανίας. Ε, η προσπάθειά μας έγινε γνωστή και σε άλλες κοινότητες. Θεωρούμε ότι είναι μια θετική αλλαγή που θα εμπνεύσει και άλλες χώρες να κάνουν το ίδιο, να υπάρξουν εκστρατείες όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά ε, να ενημερώσετε και άλλους Ευρωπαίους πολίτες ε, στις ε, δικές σας κοινωνίες ότι έχουν το δικαίωμα ψήφου. Σα Σας ευχαριστούμε πολύ για το θαυμάσιο αυτό project και νομίζω ότι σήμερα το βράδυ θα μπορέσετε να διαπιστώσετε με υπερηφάνεια ότι ο αριθμός των εκλογέων έχει αυξηθεί και μέσω της εκστρατείας σας. Ελπίζω να συνεχίσει το έργο σας αυτό και ελπίζω να βρει μιμητές και σε πολλές άλλες κοινότητες και εκτός Δανίας. Ερχόμαστε στο τρίτο βραβευμένο project Our Europe από τις κάτω χώρες. Κύριε Χέισελ, έχετε το λόγο για 7 λεπτά. Καλώς ορίσατε Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την δυνατότητα που μας δίνετε να μας παρουσιάσουμε το project μας. Περάσαμε και μερικές ε, Μερέ στις Βρυξέλλε. Γνωρίσαμε και νικητέ βραβείου, του βραβείου των προηγούμενων ετών. Πολύ σημαντική εμπειρία για μας. Σας παρουσιάσω το πρόγραμμά μας, το project μας, Are We Europe. Υπάρχει ένα μηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό στον ιστότοπό μας. Έχουμε ένα διαδραστικό ε, site ε, με διάφορες ιστορίες. Ε, είναι περισσότερο δημοσιογραφικού τύπου και λιγότερο ειδησιογραφικού τύπου. Θα ήθελα λοιπόν να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 Το βίντεο αυτό δείχνει το κίνητρό μας, για ποιο λόγο ξεκινήσαμε αυτό το project. Ε, είμαστε τέσσερις ε, φοιτητές από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Ε, έχουμε πολύ διαφορετικές σπουδές. Ο ένας είναι δημοσιογράφος, κάποιος είχε δουλέψει στο τμήμα μέσων ενημέρωσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάποιος άλλος ασχολείται με τον σχεδιασμό ιστοτόπων και είχαμε την εντύπωση ότι στα εθνικά μέσα ενημέρωσης ε, η Ευρώπη απεικονιζόταν ε, με πολύ, ε, με, με, πολύ συγκεκριμένο τρόπο, αρκετά περιορισμένο, οπότε προσπαθήσαμε παράλληλα με τα, μεταπτυχιακά μας να ξεκινήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Στην αρχή υπήρχε ένα blog στο ίντερνετ, στο οποίο διάφοροι Ευρωπαίοι πολίτες δημοσίευαν τις ιστορίες τους, και στη συνέχεια αρχίσαμε να έχουμε και ένα ηλεκτρονικό ε, ε, μηνιαίο περιοδικό στο οποίο συμμετείχαν ε, γραφίστες, σχεδιαστές ιστοτόπων και είχαμε και θεματικές ενότητες γιατί πιστεύουμε ότι η διήγηση ιστοριών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα έπρεπε να είναι απλώς ένα ντοκιμαντέρ, αλλά θα μπορούσε να συνδυαστεί με διαφόρους τρόπους ε, ε, αφήγησης των ιστοριών αυτών. Θέλαμε να δείξουμε μία διαφορετική πλευρά της Ευρώπης, διαφορετικά από αυτή που έδειχναν τα μέσα ενημέρωση στα εθνικά, να υπάρχει μία απόχρωση σε αυτήν την αρνητική παρουσίαση ε, της εικόνας της Ευρώπης, μόνο οικονομική και πολιτική. Προσπαθούσαμε να δείξουμε, να καλύψουμε αυτό το προσωπικό, το διαπροσωπικό κομμάτι της Ευρώπης που δεν είναι αρκετά εμφανές. Προσπαθήσαμε λοιπόν να υπάρχει αυτή η πανευρωπαϊκή αφήγηση ιστοριών. Ε, συνεργαζόμαστε ε, σε projects ε, τα οποία ε, αφορούν διάφορες εξελίξεις της Ευρώπης που θα διαμορφώσουν το κοινό της ε, μέλλον. Ε, ακούγονται διάφορες απόψεις, διάφορες ιστορίες που δείχνουν μια καλύτερη εικόνα του τι ακριβώς είναι η Ευρώπη. Γι' αυτό ακριβώς διαλέξαμε αυτόν τον τίτλο Are we Europe? Είμαστε η Ευρώπη για να δείξουμε ακριβώς. Ελπίζουμε να, να βρούμε μια απάντηση σε αυτήν την ερώτηση πολύ συντομότερα με τη δική μας προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Äh, Ευχαριστώ. Πραγματικά και αυτό το project είναι θαυμάσιο. Θυμούμαστε λίγο και τα έργα που βραβεύτηκαν παλαιότερα χρόνια και όταν βλέπω τον ενθουσιασμό αυτό των νέων παιδιών ε, νομίζω ότι έχουμε και το δικαίωμα να μην ανησυχούμε για το μέλλον της Ευρώπης. Βεβαίως πρέπει να γίνει και κριτική συζήτηση και να θέσουμε την ερώτηση πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την Ευρώπη που έχουμε. Ωστόσο, νομίζω ότι θα βρούμε τρόπο και δρόμο για να βελτιώσουμε πράγματι την Ευρώπη και να πείσουμε πολλούς ανθρώπους ότι ο δρόμος που ακολουθούμε είναι σωστός, λογικός και πέραν από τις διάφορες εθνικιστικές τάσεις που βλέπουμε να διαμορφώνονται εδώ και εκεί. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος δρόμος για τη στήριξη της Ευρώπης, αυτός που μας οδηγείτε εσείς. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους συντονιστές για να μπορέσουν να κάνουν παρατηρήσεις ή και ε, να θέσουν ερωτήσεις στα τρία νέα παιδιά και μετά να επανέλθω στους τρεις βραβευθέντες. Πρώτη βεβαίως η Σαμπίνε Φερχάιν. Πρώτα, ω Ευρωβουλευτή που προέρχομαι από το Ακουίσγρανον, το Άχεν δηλαδή, χαίρομαι πολύ που σα έχω κοντά μα σήμερα και που ε, ακούσαμε τα έργα σα. Νομίζω ότι το βραβείο αυτό αποτελεί και μια καλή πρωτοβουλία για να ενισχύει τον ενθουσιασμό και την δέσμευση των νέων υπέρ της Ευρώπης και να τους προσφέρει μια πλατφόρμα για να παρουσιάζουν ε, τις διάφορες πρωτοβουλίες τους, τον ενθουσιασμό τους, την δέσμευσή τους υπέρ της Ευρώπης που είναι ε, αισθητή και μέσα στην νεολαία. Ευχαριστώ όλες και όλους, όχι μόνο ε, εσάς που βραβευθήκατε, αλλά και όλες και όλους που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, γιατί υποβλήθηκαν πολλά και πολύ ενδιαφέροντα έργα, project, και είναι κάτι το οποίο προσελκύει την προσοχή μας και πραγματικά το αξίζει. έχω μια ερώτηση και προς τους τρεις σας. Τι νομίζετε ότι μπορούμε να κάνουμε εμείς από την πλευρά μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ε, υποστηρίξουμε ακόμα καλύτερα τον ενθουσιασμό των νέων. Βεβαίως κάνουμε τον αγώνα μας για να πείσουμε τις χώρες μέλη να αυξήσουν την χρηματοδότηση, αλλά πού νομίζετε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε ως ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να ενισχύσουμε τον ενθουσιασμό των νέων υπέρ της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως κυρίως το δικό σας έργο. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρος Κάμερ Εύερτ. Σίλβια Κώστα. Πολλά συγχαρητήρια για τα project τα οποία έχετε υποβάλει. Ε, εγώ ε, και από πέρσι παρακολούθησα από πολύ κοντά τη διαδικασία των βραβείων ε, Καρλομάγνου και πραγματικά η καινοτομία σας, η εφευρετικότητά σας γενικά μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εδώ βλέπουμε τους νέους τους, οι οποίοι έχουν συνηθίσει σε μια Ευρώπη χωρίς σύνορα ε, και πραγματικά όπως είπε και η νέα κοπέλα εδώ ε, μακάρι να κάνουμε μια πρόταση για 10 φορές περισσότερα κονδύλια όσον αφορά ε, το έρασμος. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που εσείς θέσατε το ζήτημα από την οπτική γωνία κάποιου που ναι μεν δεν έχει γνωρίσει την Ευρώπη με σύνορα αλλά παρόλα αυτά θέτει το ερώτημα όσον αφορά τα δικαιώματα, όσον αφορά την ίδια την ιδέα της, ε, ε, του, του τι είναι Ευρώπη και ε, εμείς που ανήκουμε στην Ευρώπη και νομίζω ότι ε, ε, πρέπει ε, πραγματικά να είμαστε συνέχεια σε επαφή με την νέα γενιά έτσι ώστε να ακούμε πώς περιγράφετε εσείς με τα δικά σας λόγια την Ευρώπη αυτό τον ανοιχτό δημοκρατικό χώρο που θεωρείται ίσως πολλές φορές σαν κάτι δεδομένο, σαν κάτι αυτονόητο. Πρέπει να δούμε τους διάφορους τρόπους έκφρασης, δημιουργίας ε, αυτούς τους τρόπους λέω που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσουμε, να επαναπροτείνουμε ε, και εν τέλει να υπεραμεινθούμε της Ευρώπης. Εμείς ε, βεβαίως συνεργαζόμαστε και με τα διάφορα φόρα και με το, ε, ε, πλατφόρμες, με το έρασμος και τα λοιπά και κάνουμε πολιτικές για τους νέους αλλά νομίζω ότι η δημιουργικότητά σας και ανοίγω παρένθεση συμφωνώ με αυτά που είπε η συνάδελφη προηγουμένως ότι θα πρέπει αυτή η δημιουργικότητα να διαχειριστεί περισσότερο προς τα μέσα ενημέρωσης τα οποία σήμερα από το πρωί συζητήσαμε έτσι ώστε να δημιουργηθεί αυτή η έννοια της κοινή ε, ε, ηθαγένειας και η ιδέα του ανήκειν ε, σε έναν κοινό χώρο. Αυτή είναι η ιδέα που έχουμε για την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κούρτσιο Μαλτέζε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, μας φέρατε έτσι έναν άνεμο ενθουσιασμού και νομίζω ότι εσείς θα πρέπει να αναλάβετε ε, ε, ε, να προωθείτε την ιδέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί η, επικοινωνία, η επικοινωνιακή πολιτική του Κοινοβουλίου δεν είναι και η καλύτερη δυνατή αυτό που με, που με ε, ενοχλεί, που με λυπεί είναι ότι τόση δημιουργικότητα από τόσους νέους χάνεται στην ουσία. Γιατί η Ευρώπη δεν έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει απασχόληση για τους νέους. Και αναρωτιέμαι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Δημοκρατία μάλιστα μπορούν να επιβιώσουν ε, όταν ε, δημιουργεί συνθήκες εργασίας ε, για τις επόμενες γενιές χειρότερες από αυτές που είχαν οι προηγούμενες γενιές. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι οι συνθήκες εργασίας των συνομιλίκων σας στις διάφορες χώρες της Ευρώπης δεν είναι καλές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σόντροβα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους εσάς. Εγώ είμαι από μια πολύ εξωτική <laughs> χώρα, είμαι από την Τσεχική Δημοκρατία ε, και πραγματικά θα ήθελα να σας εκφράσω τον σεβασμό μου. Έχω και κάποιες ερωτήσεις. Φοβόμαστε λίγο ε, για την κατάσταση στην Πολωνία και εσείς είσαστε και οι δύο από τη χώρα αυτή. Στην ερώτηση Are you Europe ε, ε, εσείς προφανώς απαντάτε θετικά. Ε, εσείς είστε νέοι και εντάσσεστε σαφώς στην προοπτική της Ευρώπης. Αλλά εσείς ως, ως Πολωνία είσαστε έτοιμοι να αγωνιστείτε έτσι ώστε να, να... να προασπίσετε την δικαιοσύνη, την ελευθερία, τη δημοκρατία γιατί στην κοινωνία σας, στις χώρες σας, ε, στην χώρα σας μάλλον υπάρχει πρόβλημα. Ε, ελοχεύουν κίνδυνοι. Σας, απο... σας ε, κάνω λοιπόν αυτή την ερώτηση και πραγματικά σας ευχαριστώ για τη δέσμευση που έχετε δείξει. Ευχαριστώ πολύ κύριο Μαλίνο. Και εγώ να σας ευχαριστήσω για τις παρουσιάσεις σας. Εγώ σε μια άλλη επιτροπή πρέπει να ψηφίσω αλλά παρόλα αυτά ε, είμαι εδώ γιατί ήθελα να σας γνωρίσω. Έπρεπε να είμαι σε άλλη επιτροπή γιατί έχουμε ψηφοφορία. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις παρουσιάσεις σας. Εγώ έρχομαι από την Βουλγαρία και εκεί προσπαθούμε να κάνουμε μια ε, φιλοευρωπαϊκή συμμαχία με έναν και μόνον στόχο στις επόμενες ε, ε, εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους νέους που θα πάνε να ψηφίσουν. Γιατί νομίζω ότι διαπιστώνεται όλοι ότι στην Ευρώπη οι νέοι όλο και πιο απομακρύνονται, δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν, απομακρύνονται από την πολιτική. Στόχος μας είναι στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές να έχουμε τις ε, εκλογές αυτές με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή νέων. Και χαίρομαι που σας ακούω σήμερα τόσο ενθουσιώδησε. Και είναι καλό να ξέρουμε ότι αυτά τα οποία γίνονται εδώ έχουν ε, αντίκτυπο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ. ναι, ναι, ο Χαίρομαι. ιδιαίτερα που είναι εδώ δύο ε, Πολωνές νικήτριες του βραβείου. Θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Έτσι λοιπόν έχω να πω ότι ε, μπράβο στους παρόντες και στις παρούσες βρίσκω ότι στα project που έχετε παρουσιάσει υπάρχει ένα κοινό στοιχείο, μια νέα προοπτική για την Ευρώπη που στρέφεται στο μέλλον, όπως είδαμε κυρίως και στο τελευταίο και τα δύο προηγούμενα project και γι' αυτό ρωτώ εσένα συνδέεται με την μελλοντική επαγγελματική σου προοπτική με την δημοσιογραφία προηγουμένως εδώ στην Επιτροπή είχαμε συζήτηση για την δημοσιογραφία στην Ευρώπη η συνειδητοποίηση για την ανάγκη προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη έχει κάποιο ε, ρόλο να παίξει και με το γεγονός που είπε ότι αισθανόμαστε καλά εντασσόμενοι και σε άλλες κοινότητες αλλού στην Ευρώπη και ποια θα είναι τα επόμενα βήματά σου. Και ερώτηση προς εσένα, ε, τις δύο ε, νέε είναι πώς θα συνεχίσετε το πρόγραμμά σας. Ευχαριστώ. Επιστρέφω τώρα το μικρόφωνο στους τρεις βραβευθέντες, μάλλον στις δύο βραβευθύσεις και τον ένα βραβευθέντα. Mm. Η κυρία Γελονίκ ας αρχίσετε εσείς πρώτοι. Καλά. Θα αρχίσω με την πρώτη ερώτηση. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει τους νέους και τις νέες να είναι πιο Ευρωπαίοι. Ποια είναι η δική μου εντύπωση. Έχουμε κάποια χρηματοδότηση για την εκπομπή μας. Εγώ έχω σπουδάσει σε διαφορετικές χώρες και βεβαίω και στην Πολωνία. Και βλέπω ότι οι νέε και οι νέοι πρώτον δεν μαθαίνουν ξένες γλώσσες. Αυτό το βρίσκω μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί κανεί να επικοινωνήσει με άλλου αν δεν μιλεί ούτε καν τα αγγλικά. Πώ θα μιλήσετε με άλλου ανθρώπου, Πώ θα συνεργαστείτε με αλλοδαπού φοιτητέ που έρχονται στην Πολωνία, α πούμε, Εκεί χρειάζεται κάποια βοήθεια. Αυτό είναι το πρώτο. Να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην εκπαίδευση. Όχι όμως για την Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικά, για τις γλώσσες. Μαθαίνοντας γλώσσες, μαθαίνει κανείς από τους άλλους. Αυτό είναι μια λύση. Όταν, όταν πήγα να σπουδάσω στην Ισπανία, οι μελέτες μου ήταν στα Ισπανικά και μιλούσα Ισπανικά. Ορισμένες φορές όταν είχαμε κάποιον στην ομάδα μας που δεν μιλούσε τα ισπανικά, το πρόσωπο αυτό έμενε εκτός. Χωρίς να θέλω να απευθύνω μομφή σε κανένα, ωστόσο, ορισμένοι πιστεύουν ότι αν κάποιος δεν μιλεί τη γλώσσα σου ή δεν μιλεί τη γλώσσα της ομάδας, είναι κάτι λιγότερο, ε, αξίζει λιγότερο το πρόσωπο αυτό. Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τις δυο πλευρές, όχι μόνο αυτούς που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα, αλλά και αυτούς που γνωρίζουν τη γλώσσα ότι θα πρέπει να είναι ανεκτική. Το άλλο είναι η εκπαίδευση στις περιφέρειες, γιατί μιλούμε για ευρωπαϊκά ε, project, για ε, εθνικά project. Εγώ έκανα το project μου μόνη μου, ήταν ατομικό. Ε, προσκαλούσα πρόσωπα, δημιούργησα την εκπομπή Πέρασα τις νύχτες μου ε, φτιάχνοντας ε, το πρόγραμμα της εκπομπής και με την τεχνική βοήθεια φίλων μου. Σε ό,τι αφορά τις πανεπιστημιακές μου σπουδές είμαι γνώμων που μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα. Αλλά, δηλαδή με τη βοήθεια του πανεπιστημίου μου. Αλλά δεν υπάρχει ένας μέντορας, ε, κάποιος δηλαδή ο οποίος να οδηγεί στα βήματά σας και να σας πει μπορείτε να κάνετε ΑΒΓ. Εγώ τέλος πάντων έχω ένα πνεύμα δημιουργικό, αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Άρα ίσως χρειαζόμαστε κάποια στήριξη. Χωρίς όμως να είναι κανείς, δηλαδή αυτός που θα σας καθοδηγήσει ο δάσκαλος, να είναι λιγότερο δάσκαλος, περισσότερο μέντορ, να σας ε, καθοδηγεί δηλαδή. Η επόμενη σας ερώτηση ήταν για την ε, ανεργία στην Ευρώπη. Αν είναι και η ερώτηση από την εξωτική χώρα. Καμιά φορά η Τσεχία είναι εξωτική χώρα. Βεβαίω αστείευτηκα. Αλλά οι Πολωνοί φοιτητέ είπαν το είπαν ως κομπλιμέντο βέβαια. Είμαστε διαφορετικοί αλλά είναι... Οι, διαφορέ διαφορές αυτές είναι καταπληκτικές και καλές. Και είναι τρελό αυτό που συμβαίνει στην Πολωνία. Και τα δύο project μας, δηλαδή το πολωνικό και το ολλανδικό, έχουν δημοσιογραφικό χαρακτήρα. Εγώ είμαι δημοσιογράφος, απαντώντας στην ερώτηση του κ. Βέντα, Σπούδασα πολιτικές επιστήμες και επικοινωνία. Όσοι δημοσιογράφοι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι για το τι λέμε στον κόσμο. Καμιά φορά και στην Πολωνία οι άνθρωποι λένε ό,τι να είναι και οι δημοσιογράφοι δηλαδή και δεν σκέπτονται ποια θα είναι η επίπτωση στο κοινό που τους ακούει αυτό το πρόβλημα είναι μεγάλο και ιδίω στην δημοσιογραφία, αλλά και στην πολιτική. Δεν βάζουν όρια ορισμένοι τι μπορούν να πούν και τι δεν επιτρέπεται να πούν. Και κάποιοι ε, φωνάζουν ή απευθύνουν κατηγορίες στους άλλους. Τώρα για την Πολωνία, δύσκολη ερώτηση και ένα πρόβλημα που αυξάνεται όχι μόνο στην Πολωνία. Εγώ το 2014 το είδα και στην Ισπανία όταν πήγα εκεί ως φοιτήτρια Έρασμος. Ίσως δεν θα έπρεπε να το πω αυτό, αλλά είναι ένα παράδειγμα. Στη διάρκεια των μαθημάτων ρώτησα την φίλη μου που μιλούσε αγγλικά μια λέξη την οποία δεν κατάλαβαινα στα ισπανικά και δεν την έβρισκα και στο διαδίκτυο, ούτε στην αυτόματη μετάφραση, ούτε στο λεξικό και ρώτησα στα αγγλικά. Και η άλλη φοιτήτρια είπε «Γιατί μιλάς αγγλικά» και απάντησα «Δεν καταλαβαίνω μια λέξη». Και μου είπε «Μην μιλάς αγγλικά, στην Ισπανία είσαι, τα Ισπανικά είναι η πιο σημαντική γλώσσα για σένα». «Μα ναι» είπα εγώ, αλλά προσπαθώ να μάθω. Και με μάλωσε και δεν κατάλαβα καλά. Μου είπε «Έρχεσαι από την Ανατολική Ευρώπη, δαπανάς ευρωπαϊκά κονδύλια και έρχεσαι εδώ για να κάνεις πλάκα». Πάντως ήταν πολύ απότομη. Θα έπρεπε να μιλάς ισπανικά. Εγώ ε, αισθάνθηκα άσχημα γιατί άρχισε ο δάσκαλος να γελά. Και τη είπα, κοίταξε, με συγχωρείς, μιλώ εκτός από τα πολωνικά και αγγλικά και γερμανικά και γαλλικά και σύντομα ισπανικά. Γιατί μου φέρες έτσι. Υπήρχε μεγάλη ανεργία στην Ισπανία τα χρόνια εκείνα και πάνω από 40% για τους νέους και ε, τους ενοχλούσε πάρα πολύ ότι έρχονταν Πολωνοί και άλλοι στην Ισπανία για να αρχίσουν να δουλεύουν. Πολλοί από τους γνωστούς μου που είχαν έρθει να σπουδάσουν έμειναν στην Ισπανία και εργάστηκαν και ορισμένοι έχουν φτιάξει και οικογένειες. Και πριν από τον ερασμό εγώ είχα πάει και μάζευα στα φίλια και ήμασταν Ισπανοί και Πολωνοί και δουλεύαμε μαζί. Εμεί νέοι και νέε δεν μπορούσαμε να βρούμε άλλη δουλειά στι χώρε μα. Ολοκληρώστε τώρα, λέει η Πέτρα. Για το μέλλον. Αυτό που θα ήθελα να κάνω στο μέλλον έχει βέβαια σχέση με τις σπουδέ μου. Εγώ εργάζομαι σε γραφείο σύνταξης στην Πολωνία. Θέλω να δουλέψω στο ραδιόφωνο. Σήμερα μαγνητοφωνήσαμε εκπομπή, μάλλον ε, ε, ναι, μαγνητοφωνήσαμε εκπομπή για το ραδιόφωνο εδώ. Ε, εγώ δεν είμαι φοιτητή πλέον, άρα δεν μπορώ να δουλέψω πλέον στον φοιτητικό ραδιοφωνικό σταθμό. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να δουλέψω σε ένα μεγαλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό. Υπάρχουν και άλλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί των φοιτητών. Ράδιο Ράκτα τη Σόφια, τη Σόφια δηλαδή στη Βουλγαρία και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί είναι και στα αγγλικά μάλιστα και μπορείτε να το ακούσετε και αλλού και ε, μάλιστα εκπέμπει και σε όλη την Ευρώπη. Και είμαι πολύ ικανοποιημένη για αυτό το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λέει η Πέτρα Κάμερ Εύερτ. Εσείς τώρα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Εσείς ε, ως Κοινοβούλιο, ως Ευρωπαίοι Βουλευτές, τι μπορείτε να κάνετε για τα project μας. Μίλησα προηγουμένως ε, για το δικαίωμα ψήφου. Σε λίγο, όχι πολύ, ε, σε πολύ χρονικό διάστημα θα έχουμε τις ευρωπαϊκές εκλογές. Μπορείτε να μιλήσετε ε, στις χώρες σας σε Ευρωπαίους πολίτες που περιμένουν να ακούσουν για την Ευρώπη. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν φωνή, δεν ακούγεται η φωνή τους και που πρέπει και θέλουν να ακουστεί η φωνή τους. Υπάρχει ένα έλλειμμα δημοκρατίας ε, κατά αυτή την έννοια ε, στα ευρωπαϊκά όργανα και εγώ βλέπω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν ε, σημείο διασύνδεσης, σαν δυνατότητα διασύνδεσης των πολιτών με τα όργανα τα ευρωπαϊκά και το θέμα της εκμάθησης γλωσσών είναι σημαντικό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ίσως και να ταξιδεύουν, ίσως και να βγαίνουν από, τη χώρα τους, αλλά δεν μιλούν ε, ξένες ε, γλώσσες ε, και είναι ένα πρόβλημα σχετικά με το τι συμβαίνει στην Πολωνία, μια και είμαι πολωνικής καταγωγής. Ε, κοιτάξτε, Νομίζω ότι πρέπει κανείς να προχωράει με μικρά βηματάκια. Ε, η οικογένειά μου είναι πολύ συντηρητική. Έχω την αίσθηση ότι κάθε φορά είναι σαν ένα μωρό που ε, κάνει τα πρώτα του βήματα. Ε, προσπαθώ να τους μεταφέρω κάποια πράγματα. Και όμως κάθε φορά που επιστρέφω στην Πολωνία έχω την αίσθηση ότι ξαναρχίζουμε από την αρχή είναι σημαντικό ε, στις ε, χώρες της Ευρώπης και προκειμένου η Πολωνία είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα ε, να υπάρχει δημοκρατία, να υπάρχει δυνατότητα για όλους να εκφραστούν σχετικά με την εκστρατεία για το δικαίωμα ψήφου. Να σας πω ότι έχω ένα φίλο που είναι εκπρόσωπος της νεολαίας σε, περιφερειακά, σε περιφερειακών οργάνων και εκεί ε, πρέπει να εξηγήσουμε όπως και σε, εθνικό επίπεδο και σε περιφερειακό το τι ε, συμβαίνει ε, να σας πω ότι μας βοήθησε αυτό, η συμμετοχή του σε αυτό το όργανο να κάνουμε μια μικρή εκστρατεία για την ψήφο και στην Δανία. Νομίζω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να, να κάνετε εκστρατεία προς όλους όσοι κατοικούν στη χώρα σας, όχι μόνο σε αυτούς που μιλούν τη γλώσσα σας. Ο επόμενος παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ για τα ενθαρρυντικά λόγια και τις ερωτήσεις που υποβάλλατε σχετικά με το πώς μπορούμε να εμπλέξουμε περισσότερο τους νέους νομίζω ότι είναι καλό να πούμε ότι ήδη συμβαίνουν αρκετά πράγματα, υπάρχουν αρκετά ε, ευρωπαϊκά projects για τους νέους που τρέχουν ήδη και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και πρέπει να συνεχίσουν αλλά για να είμαι ειλικρινή, ε, αν δείτε ποιοι συμμετέχουν στα ε, project αυτά, είναι νέοι με υψηλά προσόντα, με μεγάλο βαθμό εκπαίδευση, ας πούμε, θα πρέπει να υπάρξουν προγράμματα για ανθρώπους ε, που έχουν ε, δυσκολία να βρουν δουλειά, που είναι στο περιθώριο, που είναι άνεργοι και βεβαίως και ε, ε, νέους στον ε, τομέα τον δημιουργικό είτε είναι δημοσιογράφοι φυσικά αλλά και στον δημιουργικό, στους καλλιτέχνες κλπ. Εκεί μιλάμε για έναν ιδιαίτερα σταθή κλάδο και όταν οι άνθρωποι αυτοί καταφέρνουν να συνενωθούν και να δουλέψουν μαζί μπορεί να κάνουν εκπληκτικά πράγματα. αυτό είναι ένα πεδίο ας πούμε ε, που ε, θα θέλαμε εμείς ε, να συμβάλλουμε με την πλατφόρμα μας αλλά πολλά περισσότερα μπορούν να γίνουν. Επίσης το πρόγραμμα Εράσμους αφορά κυρίως τους πανεπιστημιακούς φοιτητές υπάρχουν όμως και οι νέοι οι οποίοι έχουν πιο πρακτική εκπαίδευση και αυτοί οι άνθρωποι ίσως δεν έχουν τόσο μεγάλη ε, εμπειρία, δεν έχουν ε, δεν έχουν τις εμπειρίες ε, που έχουν οι νέοι οι οποίοι πηγαίνουν σε άλλες χώρες με το αέρασμος. Εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι θα πρέπει να διευρυνθεί ο κύκλος των νέων που εντάσσονται σε projects. Όσον αφορά το μέλλον, πολύ δυναμικό υπάρχει στο μέλλον. Εμεί θα θέλαμε να αναπτύξουμε την πλατφόρμα ε, και να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε με άλλες ε, ε, αντίστοιχες πλατφόρμες. Και καλό είναι γενικά να μην σκέφτεται κανεί μόνο το δικό του project, τη δικιά του πλατφόρμα, αλλά να συνεργάζεται, να ανοίγεται σε άλλες, έτσι ώστε να βρεθούν τρόποι ώστε να δημιουργούνται ψυχολογικά βέβαια και πολιτιστικά ε, αγαθά αλλά ε, και γενικότερα στοιχεία τα οποία θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν όλοι για ανάπτυξη εμπορικών, ε, πολιτιστικών προγραμμάτων, αγαθών κτλ πολλά συμβαίνουν, μεγάλη δημιουργικότητα υπάρχει, αλλά νομίζω ότι το σημαντικό είναι ο ένας να μάθει από τον άλλον, έτσι ώστε ε, στο μέλλον η κατάσταση να είναι πολύ καλύτερη. Αυτά νομίζω ότι απήντησα στις ερωτήσεις σας. Α, όσον αφορά την ενεργεία, Βεβαίως σε μερικές χώρες η ενεργεία είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε ε, άλλες. Δεν έχω φυσικά μια έτοιμη λύση, έστω και αν έχω σπουδάσει οικονομικά Η αίσθησή μου είναι ότι πρέπει να βρούμε λύσεις, ε, όχι μόνο μέσω της μετανάστευσης λοιπά. Νομίζω ότι είναι καλό οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν ε, να ε, μετακινούνται από τη μία χώρα στην άλλη όταν η χώρα στην οποία βρίσκονται δεν έχει πολύ οικονομική, αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, αλλά το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι και απέναντι στη μετανάστευση η Ευρώπη να παραμείνει ε, ενωμένη και να καταλάβει ότι και στην μετανάστευση μπορεί να βρει μια νέα δύναμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς τώρα πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ την ε, συζήτηση και λυπούμε πολύ, αλλά σας ευχαριστώ που περάσατε σήμερα από εδώ και παρουσιάσατε το έργο σας ε, αντιληφθήκατε ότι όλοι εδώ είναι ενθουσιασμένοι από τη δέσμευσή σας. Ελπίζουμε να συνεχίσετε αυτά που κάνετε και με νέες ιδέες και με νέα project. Η ανταλλαγή απόψεων ε, που είχατε εδώ για ένα διήμερο στις Βρυξέλλες και με άλλους βραβευθέντες από παλαιότερα έτη, ίσως ε, προκύψουν και νέες ιδέες από αυτό και να δημιουργηθεί ένα είδος ε, ντόμινο effect το οποίο να μας επιτρέψει να προχωρήσουμε μερικά βήματα παραπέρα. Να συζητούμε τα προβλήματα όπως πραγματικά εμφανίζονται και σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ που ήλθατε στις Βρυξέλλες και σας εύχομαι να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες και ημέρες. Καλώ συνεχίζει η πρόεδρο, τώρα θα πρέπει να συνεχίσουμε την ημερήσια διαταξή μα. Η Χέλγκα τα κατάφερε να φτάσει, η κυρία Τρίπελ. Να πω για το πρώτο τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης για την έκθεση του Κόρτσιο Μαλτέζε. Η προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών είναι 30 δεκάτου στι 2 το απόγευμα. Θα σας το στείλω και γραπτός, αλλά θα ήθελα να σας το πω και προφορικός. 30 ενδεκάτου 14.00. Μας μένουν 7 λεπτά για την εξέταση. Όχι. Λάθος ε, φάκελος για το σώμα αλληλεγγύης και μιλώ για την εξέταση των τροπολογιών. Έλγα, σου παραδίδω μέσω στο μικρόφωνο για να μπορέσεις να μας πεις λίγα λόγια και ιδίως πόσες τροπολογίες έχουν φτάσει στο γραφείο σου και πώς θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Just in time. Ε, χρειάστηκε να... να βρω άλλες ε, ε πτήσεις, διότι 5,5 ώρα που έφτασα εκεί είχαν ήδη κλείσει την ε, θηρίδα. Έχουμε 600 τροπολογίες τώρα, μα ίσως όχι και πάρα πολλές. Ε, πολλές πάντως τις υποστηρίζει η Επιτροπή Καλτ. Η κυρία Μπίλδη και ορισμένοι άλλοι από τα δεξιά κόμματα που είναι αντίθετοι με την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη διότι τους μυρίζει πολύ η Ευρώπη, οι υπόλοιποι υποστηρίζουν λίγο πολύ τα όσα προτείνω. Δηλαδή, η πλειοψηφία είναι υπέρ της αλλαγής του ονόματος να πάψει να λέγεται σώμα και να λέγεται πρωτοβουλία, πιο ξεκάθαρο, μου αρέσει και το υποστηρίζω. Το ίδιο σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής περιοριστεί ιδίω σε νέους, σε νεολαία η οποία ε, βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, σαφής πλειοψηφία να αρχίσουμε από τα 18 χρόνια και να μην κατέβουμε στα 16, διότι δεν είναι ενήλικα τα πρόσωπα αυτά και δεν μπορούν να υπογράφουν συμβάσεις χωρίς τους γονείς τους και ούτε μπορούν να μεταβαίνουν αλλού στην Ευρώπη ή αλλού για να πάμε και παραπέρα δηλαδή εκτός από τις 28 χώρες μέλη, αλλά να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στι γειτονικέ χώρες, αυτό που θέλουμε δηλαδή ως common line, γιατί θέλουμε περισσότερη αλληλεγγύη και ιδίω προ την Ανατολική Ευρώπη. Και υπάρχει και μια σαφή ε, πλειοψηφία κατά του occupational trend και για να πω χρήμα. Όλοι δηλαδή και εσείς και εγώ θέλουμε φρέσκο χρήμα. Καλώς έχουν λοιπόν οι τροπολογίες από τη δική μου σκοπιά οι πιο εύκολες τροπολογίες που έχω λάβει εδώ και 13 χρόνια που, βρίσκομαι, που είμαι ευρωβουλευτής, ας προχωρήσουμε και νομίζω θα επιτύχουμε μια ευρεία πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ αγαπητή Χέλγκα, γιατί παραπονιόμουν το πρωί δεν έχουμε καμιά φορά και κανένα θέμα απλό και εύκολο. Αν έχετε πλειοψηφία είναι εύκολα τα πράγματα λέει η κυρία Τρούπελ. Φαίνεται πως αυτό συμβαίνει στην περίπτωσή σου και φαίνεται πως συμφωνούμε όλοι οι περισσότεροι έχουμε άλλο χρόνο τέσσερα λεπτά άρα ένα λεπτό για τον καθένα γιατί ακριβώς 11.30 πρέπει να αρχίσουμε την συνεδρία των συντονιστών Σόιντροβα Μάλιστα, ομιλία ενός λεπτού δηλαδή με άλλα λόγια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εισαγωγή στο θέμα. Όντως είναι πολλές οι τροπολογίες. Ο στόχος μας θα είναι να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε επί συμβαστικών τροπολογιών και η πρώτη θα πρέπει να είναι για την ίδια την ονομασία. Τονίζω ότι στόχος μας θα πρέπει να είναι να δώσουμε έμφαση στον χαρακτήρα πρωτοβουλίας Θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη ε, έμφαση λοιπόν στον πρωτοβουλιακό χαρακτήρα. Η Επιτροπή Απασχόλησης θα επιμείνει νομίζω στο να διατηρηθεί ο επαγγελματικός χαρακτήρας. Θα πρέπει εμείς λοιπόν να σκεφτούμε τι θα κάνουμε στην περίπτωση αυτή. Σίλβια. Ευχαριστώ πολύ, Χάλικα Τρούπερ, για την τοποθέτηση που έχει απέναντι στην πρόταση. Μονάχα μερικά σημαντικά σημεία. Να πω ότι συμφωνώ λοιπόν και το ξεκαθαρίσαμε με τις τροπολογίες μας, η έναση του τι σημαίνει ε, εθελοντική, εθελοντισμός, εθελοντική σχέση και αλληλεγγύη. Δεύτερον, ότι θα πρέπει να είναι δημόσια και οι ε, οργανώσεις πρέπει να είναι δημόσιες και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Και τρίτον, ε, να υπάρχουν αποζημιώσεις επιστροφές ε, ε, εξόδων και επίσης να ε, ε, εξακολουθούν να, υπάρξουν, να ε, υπάρχουν οι λεγόμενες sending organizations. Εγώ, εσύ το λες ενδιάμεσο. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει οπωσδήποτε να, υπάρχουν, να υπάρχει παρακολούθηση όσον αφορά την αρχική φάση, την κατάρτιση κτλ. Και όλες οι οργανώσεις οι οποίες, δηλαδή να το πω διαφορετικά, θα πρέπει να υπάρχει το πόρτο, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν και αυτές οι συνοδευτικές. Επίσης να ε, σας πω ότι ξέρετε τι συνέβη στο Συμβούλιο Υπουργών ε, όσον αφορά τα, τις δαπάνες, όσον αφορά τα χρήματα κτλ. Η κυρία Χιμένερ. Πολύ σύντομα ευχαριστούμε Μεχέλγα για την δουλειά που έκανες. Πολύ μου αρέσει η ιδέα της ε, πρωτοβουλίας. Εγώ είχα προτείνει την λέξη δράσης, action, όσον αφορά την αντικατάσταση του σώματος. Η συζήτηση για τον συνδυασμό των δύο στελεχών, των δύο τμήματων της πρωτοβουλίας θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι έχουμε συμφωνήσει σε αυτό. Ε, όσον αφορά το δημοσιονομικό, πιστεύω ότι θα πρέπει ε, να εξακολουθήσει η χρηματοδότηση του Erasmus ε, Plus αλλά θα πρέπει να ζητηθεί και η γνώμη της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμών όσον αφορά το θέμα αυτό. όχι μόνο τα κράτη-μέλη αλλά και άλλοι μπορούν να συμμετάσχουν. Εγώ είμαι υπέρ αυτή τη άποψη και ε, γενικά πιστεύω ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό πρόγραμμα για να προωθηθούν ιδέε οι οποίε είναι πραγματικά βασικέ για μα. Ευχαριστώ. Τέλο, ο κύριο Μαλτέζη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, για την εξαιρετική εργασία. Οποιοδήποτε γνωρίζει ε, τις εθελοντικές οργανώσεις, ε, ξέρει ότι υπάρχει αυτή η πρακτική των επιστροφών των αποζημιώσεων για τις αποστολές. Ε, και ξέρετε ότι ε, όλες αυτές οι κινήσεις έχουν πάρα πολύ και οι συμμετοχές ε, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό σύν ακόμα και για την επαγγελματική διαδρομή των νέων. Επίσης τους δίνει τη δυνατότητα να συνεργαστούν, να λύσουν από κοινού προβλήματα και αυτό στην, σε μια οργανωμένη κοινωνία αποτελεί μεγάλο προτέρημα και μεγάλο προσόν. Επομένως, αυτές οι εθελοντικές οργανώσεις μπορεί να αποδειχθούν πολύ χρήσιμες ε, για την μετέπειτα επαγγελματική ζωή. Αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσουμε τον αθλητικό χαρακτήρα και η ελληνική θα πρέπει να παραμείνει ε, δωρεάν ε, γιατί πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική ανθρώπινη αξία. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε τον Πάπα μονάχο του να παίζει σε αυτό το, το πεδίο. Επομένω, εγώ επιμένω ότι η αλληλεγγύη πρέπει να δίνεται δωρεάν. Θα πρέπει να βρούμε μια σωστή μέση λύση, ένα σωστό συμβιβασμό weiteren Wortmeldungen mehr zulassen. Alles Weitere muss dann in den Schattenberichterstattertreffen diskutiert werden oder am Rande. Wir haben einfach die Zeit nicht mehr, Helga noch. Only one additional information. The shadow meetings on the 30th of November together with EMPL, so we will have maybe, then we will know more what EMPL is going to do and what about the majorities. Here the majority is clear, in EMPL it's open, so far as I know. We will see.